ελπίζουμε να μπορέσουμε όλοι μαζί να επιτύχουμε τους στόχους μας και να καταλήξουν οι διαπραγματεύσεις πριν λήξει ο χρόνος. Κυρίε και κύριοι συνάδελφοι, έλαβα μία πρόταση ψηφίσματος για την ε, συζήτηση αυτή, για το θέμα της συζήτησης αυτής. Έληξε η συζήτησή μας και η ψηφοφορία θα διεξαχθεί σήμερα το μεσημέρι στις 12 η ώρα δηλαδή. Τώρα ερχόμαστε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης που είναι κοινή συζήτηση σχετικά με την Ευρώπη 2020, κατευθυντήριες γραμμές για την πολιτική απασχόληση. Έχουμε τις δηλώσεις του Συμβουλίου και της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής και έχουμε την έκθεση Μπέρες ε, που αφορά τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών και τη δήλωση της Επιτροπής για την εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών για την πολιτική των κρατών μελών στον τομέα της ε, απασχόλησης. Ε, ξεκινούμε τη συζήτηση με τον Υπουργό, τον κύριο Μαρτώνη, εξ ονόματος του Συμβουλίου. Mr. you have the Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, καλωσορίζω ιδιαίτερα την ευκαιρία αυτή για να μιλήσω ενώπιον σας για ένα θέμα πολύ σημαντικό για την Ουγγρική Προεδρία. Την στρατηγική για την Ευρώπη του 2020 που είναι πολύ σημαντικό θέμα για όλους μας μάλιστα. Είναι σαφές ότι η Ευρώπη πρέπει να ξεπεράσει μια σειρά σοβαρών προκλήσεων εάν θέλει να παραμείνει ανταγωνιστική με τον υπόλοιπο κόσμο. Κάποιες από τις προκλήσεις αυτές προκλήθηκαν από την χρηματοοικονομική και οικονομική κρίση. Κάποιες από αυτές ωστόσο είναι εγγενείς στην, ε, στην μικρή αποφασιστικότητα και τις, περι, τους περιορισμένες δυνατότητες που έχουμε να καλύψουμε και να τηρήσουμε τις, τους στόχους της στρατηγικής της Λισαβόνας. Όπως συχνά αναφερθήκε, μια κρίση μπορεί να είναι και μια ευκαιρία και στα αρχαία ελληνικά και στα κινέζικα η έννοια κρίση μπορεί να σημαίνει λύση εν ώψη, μια πορεία προς τη λύση. Γι' αυτό το λόγο πιστεύουμε ότι η κρίση είναι βασικός παράγοντας παρέχοντας κίνητρα και παρατρύνοντας τα κράτη-μέλη να υιοθετήσουν μια νέα ευρωπαϊκή στρατηγική για θέση εργασίας και έξυπνη και βιώσιμη ανάπτυξη. Αυτό είναι, αυτά είναι τα χαρακτηριστικά της στρατηγικής Ευρώπη 2020. Ε, πιστεύουμε ότι η στρατηγική αυτή θα βοηθήσει την Ευρώπη να, να κάμψει από την κρίση και να γίνει ισχυρότερη και εσωτερικά και σε διεθνές επίπεδο προωθώντας την παραγωγικότητα, την ανάπτυξη την κοινωνική συνοχή και την οικονομική διακυβέρνηση. Όλα αυτά είναι αναγκαία εάν θέλουμε να παραμείνουμε ανταγωνιστικοί σε παγκόσμιο επίπεδο, ιδίω εν ώψη τη αύξηση, τη σημαντική αύξηση των αγορών τη Ασία. Επίση είναι ουσιαστικό κάτι τέτοιο για να διαφυλάξουμε το κοινωνικό μοντέλο, τον τρόπο ζωή μα, που είναι βασικό χαρακτηριστικό τη Ευρώπη, που ενστερνιζόμαστε και που πρέπει να διαφυλάξουμε. Η στρατηγική του 2020 επιβεβαίωσε πέντε βασικούς στόχους της Ένωσης που είναι κοινή στόχοι στις δράσεις των κρατών μελών και της Ένωσης. Βελτίωση συνθήκων ζωής, προώθηση της ε, ανάπτυξης, ε, κάλυψη των ε, στόχων αλλαγής κλίματος και ενέργειας, βελτιώνοντας τα επίπεδα εκπαίδευση και προωθώντας την κοινωνική συνοχή ιδίως μέσω της μείωσης της φτώχειας. Ως τμήμα της επίτευξης των στόχων αυτών η Επιτροπή ε, παρουσίασε επτά βασικές πρωτοβουλίες με τις δράσεις που προτείνει να λάβει για την ενίσχυση της ενίας αγοράς και την παρότρινση της ανάπτυξης και, της, ε, και των θέσεων εργασίας. Ψηφιοποίηση, κινητικότητα νέων, αποφασιστική πολιτική εκβιομηχάνησης, ατζέντα για νέα προσόντα και νέες θέσεις εργασία και μια ευρωπαϊκή πλατφόρμα κατά της φτώχειας. Κάθε μία από τις πρωτοβουλίες αυτές σημαίνει ότι πρέπει να υπάρξει συντονισμός ένωσης και κρατών μελών, ούτω ώστε οι δράσει σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο να ενισχύουν η μία την άλλη. Το Δεκέμβριο του 2010, η πρώτη έκθεση υλοποίησης της που προετοίμασε η Προεδρία σε συνεργασία με την Επιτροπή και την επερχόμενη Ουγγρική Προεδρία έδωσε μια γενική επισκόπηση των εργασιών ε, που ξεκίνησε με την στρατηγική του περασμένου Ιούνιο. Το κείμενο αυτό υπογραμμίζει τις σημαντικές, σημαντικότερες δουλειές ε, στα διάφορες, στις διάφορες συνθέσεις του Συμβουλίου για τις 7 πρωτοβουλίες που ανέφερα. Ενώ αναγνωρίζει και διαπιστώνει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί σε διάφορους τομείς πολιτικής και που παίζουν σημαντικό ρόλο στην συνολική στρατηγική. Ενιαία αγορά, πολιτική συνοχής και γεωργία ταυτόχρονα παριθμεί τι δραστηριότητε και των πρωτοβουλειών ε, και τις πρωτοβουλίες που έχουν διεξαχθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο το τελευταίο εξάμεινο για του πέντε βασικούς στόχου της Ένωσης. Θέλω να υπογραμμίσω κάποια σημαντικά στοιχεία για την οικονομική διακυβέρνηση τώρα. Η εφαρμογή της οικονομικής της μεταρρύθμιση στην οικονομική διακυβέρνηση είναι θεμελιώδης προπόθεση για την αντιμετώπιση της κρίσης και την ενίσχυση της ευρωπαϊκής οικονομίας. Γι' αυτό το λόγο η στρατηγική του 2020 συνδέεται στενά με το λεγόμενο ευρωπαϊκό εξάμεινο. Βασικό εργαλείο για μακροοικονομική εποπτεία που θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά υπό την Προεδρία μας. Η διαδικασία αυτή ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2011 με την παρουσίαση των ετησίων, ε, της έρευνας για την ανάπτυξη της Επιτροπής. Η Ουγγλική Προεδρία ε, δίνει ιδιαίτερη προσοχή στην διασφάλιση ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο θα προχωρήσει ε, επιτυχώς και χωρίς προβλήματα. Και για το σκοπό αυτό θα οργανώσουμε μια σειρά συζητήσεων σε όλες τις συνθέσεις του Συμβουλίου εν ώψη του, Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Μαρτίου. Το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων ε, θα αναλάβει ε, μια συνθετική έκθεση για την συνάντησή της, 21, τη συνάντησή της 21 Μαρτίου που θα περιλάβει τα βασικά μηνύματα των εργασιών που έχουν, ε, που έχουν ολοκληρωθεί σε διάφορα συμβούλια. Η έκθεση αυτή θα υποβληθεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μαρτίου και θα αποτελέσει τη βάση των σχετικών συζητήσεων με στόχο την συμφωνία μια σειράς επί μια σειράς προτεραιοτήτων για διαρθρωτικές και ε, ε, ε, ε, και, δημοσιονομική, και δημοσιονομική διασφάλιση. Επίσης τα κράτη-μέλη θα εξασφαλίσουν ότι θα ετοιμάσουν εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεις και προγράμματα σταθεροποίησης που θα υποβάλουν τον Απρίλιο στην Επιτροπή. Κατόπιν θα συνεχιστεί η δουλειά για την επεξεργασία συγκεκριμένων συστάσεων προς συγκεκριμένα κράτη-μέλη που θα ληφθούν υπόψη από τα κράτη-μέλη όταν ολοκληρωθεί ο προπολογισμό των χωρών αυτών για το 2012 και όταν υλοποιούν τις στρατηγικές ανάπτυξης τους. Αναγνωρίζω ότι το χρονοδιάγραμμα αυτό είναι πιεστικό. Ωστόσο, πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τον Ιούνιο-Ιούλιο. Κύριε Πρόεδρε, κυρία, κυρίες και κύριοι βουλευτές, η στρατηγική Ευρώπη 2020 είναι βασική για να διασφαλίσει την μελλοντική οικονομική επιτυχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνδέεται στενά με τις μεταρρυθμίσεις στην οικονομική διακυβέρνηση που επίσης θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο. Για να μείνουμε ανταγωνιστικοί και να εξασφαλίσουμε ανάπτυξη στο μέλλον, Αλλιώ δεν θα μπορέσουμε να διατηρήσουμε και υψηλό επίπεδο κοινωνική προστασία στο εσωτερικό μα και να προωθήσουμε τον ρόλο τη Ευρώπη προ τα έξω. Αυτό αποτελεί μια σημαντική πρόκληση για τα επερχόμενα έτη στην Ευρώπη και είμαι βέβαιο ότι θα, λάβω... θα λάβουμε την υποστήριξη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην επιτυχία των στόχων αυτών. Ευχαριστώ. Thank you, ευχαριστούμε κύριε Προεδρεύοντα για την εισαγωγή σας αυτή. Κάνουμε λόγο για ένα πολύ σημαντικό θέμα, τη στρατηγική για την Ευρώπη του 2020 και έχουμε και ένα πολύ υψηλό ποσοστό ανεργίας. Η μεγαλύτερη αυτή υπόθεση, η πολιτική δηλαδή για την απασχόληση, έχει κέρια σημασία και για την στρατηγική μας και ο αρμόδιος επίτροπος ο κύριος Λάσλο Άντορ εξ ονόματο τη Επιτροπής. Καλώς ήρθατε στο Κοινοβούλιο, θα λάβει τον λόγο. Έχετε τον λόγο κύριε Επίτροπε, σα ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ κύριε, Επίτροπε, κύριε Προεδρεύοντα Μάτων. Όπω γνωρίζετε έχει υιοθετήσει την πρώτη ε, η, ε, ε, έκθεσή τη η Επιτροπή για την στρατηγική αυτή είναι ε, μια νέα εκκίνηση σε σχέση με το παρελθόν και ένας νέος συντονισμός για αυτό το εξάμεινο. Η κύρια ιδέα για αυτό το ευρωπαϊκό εξάμεινο είναι πολύ απλή. Να διασφαλίσουμε τη σταθερότητα της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Δεν έχουμε άλλη επιλογή παρά να κάνουμε έναν εξάντε συντονισμό, έναν εκπροημίου συντονισμό μεταξύ των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα αίτια της κρίσης σε κάποιες χώρες της ε, ΟΝΕ καταδεικνύουν αυτό ε, πρόδειλα. Και δείχνουν όλα αυτά ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει πόσο στενά συνδέονται οι οικονομίες των κρατών μελών και πώς οι πολιτικές σε ένα κράτος μέλος μπορεί να έχουν επιπτώσεις σε ένα άλλο και η διαχείριση του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου θα είναι μια δοκιμασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση, μια λιδία λίθος. Θα πρέπει να δούμε και τις εταιρικέ σχέσεις που αποτελούν ε, ιδιαίτερο, έχουν ιδιαίτερο ρόλο για μας θα πρέπει να αποδειχθεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να ταυτοποιήσει τις ε, μεταρρυθμίσεις εκείνες συνολικά που είναι οι πιο κατεπίγουσες και να δώσει τις σωστές πολιτικές απαντήσεις. Η αιτήσια αυτή αναθεώρηση είναι σαφής ε, στις προτεραιότητες. Μία ολοκληρωμένη προσέγγιση υιοθετεί για τις κύριες δράσεις ε, που πρέπει να γίνουν υπό τρία κεφάλαια, υπό τρεις άξονες. Πρώτον, μια παγίωση των δημοσιονομικών και εξυγίανση και αναδιάρθρωση του ε, οικονομικού τομέα για την μακροοικονομική σταθερότητα δεύτερον μεταρρυθμίσεις διαρθρωτικές ε, για μεγαλύτερη απασχόληση και μέτρα τα οποία θα δώσουν δυνατότητα ανάκαψης ε, Ελήφθησαν υπόψη τα κύρια μελήματα για αυτή την αναθεώρηση και φαίνεται ότι ε, θα υπήρχε ίσως κάποια παρέκκληση από τις ε, ολοκληρωμένες αρχές. Όμως θέλω να είμαι σαφής επ' αυτού. Επέλεξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εστιάζεται σε αυτή την αναθεώρηση για να, την ρύθμιση των πιο κατεπηγουσών αναγκών και για τις μεταρρυθμίσεις εκείνες που είναι αναγκαίες για την οικονομική ανάκαμψη και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Η ετήσια αυτή έκθεση είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη με τις κατευθυντήριες γραμμές και για την απασχόληση. Καλωσορίζουμε την υποστήριξη του Ευρωκοινοβουλίου στις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να παραμείνουν οι κατευθυντήριες γραμμές αναλύωτες για το 2011. Είναι σημαντική αρχή να διασφαλιστεί ένα σταθερό πλαίσιο για αυτές τις στρατηγικές μέχρι το 2014 ώστε τα κρατη να έχουν επαρκή χρόνο να υλοποιήσουν τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις. Οι κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση και αυτές αποτελούν βάση αυτής της ετήσιας έκθεσης που ταυτοποιούν τα πιο αναγκαία μέτρα και τα πιο κατεπήγοντα μέτρα για την απασχόληση. Πρώτον, την εισαγωγή συστημάτων φορολόγησης μεταθέτοντας το βάρος της φορολογίας από τους μισθούς σε άλλα πεδία. Δεύτερον, να υπάρξει η δυνατότητα ανακούφισης όσον αφορά το βάρος το οικονομικό της ε, φορολόγησης και να υπάρχει η δυνατότητα ανάπτυξης οικονομικής με θέσεις απασχόλησης ώστε να μπορέσουν οι πολίτες να ε, ενεργοποιηθούν και να αυτοαπασχοληθούν όπου γίνεται και να υπάρξει δυνατότητα και οι κατευθυντήριες γραμμές θα αποτελέσουν τη βάση για συγκεκριμένα μέτρα όσον αφορά συγκεκριμένα κράτη ώστε θα με βάση το άρθρο 148 της συνθήκης να μπορέσει να λειτουργήσει αυτή η πρωτοβουλία. Είναι βάση αυτή η ετήσια έκθεση για την συζήτηση και τις κατευθυντήριες γραμμές που θα πρέπει να ακολουθηθούν από τα κράτη-μέλη προσδοκά ότι τα κράτη-μέλη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσδοκά ότι τα κράτη-μέλη θα αναλάβουν πρωτοβουλίε για την υλοποίηση αυτών των κατευθυντήριων γραμμών και με τα εθνικά προγράμματα που θα ευθυγραμμιστούν με τη στρατηγική για την Ευρώπη του 2020 θα εξεταστούν αυτά κατά το δεύτερο μέρος του Απριλίου και με βάση αυτή την εξέταση και ευθυγραμμιζόμενοι με τι υποχρεώσει των συνθηκών θα προτείνουμε συγκεκριμένες κατευθυντήριε γραμμέ για κράτη-μέλη που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και θα ολοκληρωθεί και ο προπολογισμό για το 2012. Οι κατευθυντήριε γραμμές για τις πολιτικές θα πρέπει να υιοθετηθούν από το Συμβούλιο πριν από το καλοκαίρι. Πρόεδρε, αξιότιμοι Ευρωβουλευτέ, θα ήθελα να ολοκληρώσω τονίζοντα τη σημασία του ρόλου σα για την επιτυχή έκβαση της στρατηγικής για την Ευρώπη του 2020 ιδιαίτερα όσον αφορά αυτές τις πρωτοβουλίες ο ρόλο σας ως συνομοθέτη είναι πολύ σημαντικό. θα πρέπει να, να δημιουργηθούν οι αναγκαίες θετικές εκείνες προϋποθέσεις για την επίτευξη αυτών των στόχων η συζήτηση των πολιετών δημοσιονομικών προοπτικών θα ξεκινήσει σύντομα. Υποβάλλει τις προτάσεις της μέχρι τον Ιούνιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο ρόλος σας ως δημοσιονομικού σκέλους θα είναι κέριος για να διασφαλιστεί η πολιτική για το 2020 και των προτεραιοτήτων που θα πρέπει να αντανακλώνται στον προϋπολογισμό. Αν θέλουμε να είμαστε αξιόπιστοι θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα ευθυγραμμίζονται αυτές οι προτεραιότητες με τις πολιτικές που θα υιοθετήσουμε και τις ε, μεθόδους για την επίτευξή τους. Είναι περισσότερο αναγκαίο από ποτέ να δείξουμε ότι αυτή η προσπάθεια θα δώσει μια πρόσθετη αξία και ότι αυτή η συντονισμένη προσπάθεια θα μπορεί να δώσει καλύτερο αποτέλεσμα από ότι οι εθνικές ε, επιμέρους προσεγγίσεις. Θα πρέπει λοιπόν να δραστηριοθούμε σε όλα τα επίπεδα. Μόνο όταν όλοι διαδραματίσουν το ρόλο τους στην επίτευξη αυτών των στόχων και ακολουθηθεί η σωστή πορεία θα μπορέσουμε να είμαστε επιτυχείς. Ευχαριστώ. Uh, και εγώ σας ευχαριστώ. Επόμενη ομιλήτρια είναι η συγγήτρια, η κυρία Περβάνς και Μπερές. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Προεδρεύοντα του Συμβουλίου, κύριε Επίτροπε, εξ ονόματος της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων και Απασχόλησης, Χαίρομαι ιδιαίτερα για την πρώτη αυτή ευκαιρία που έχουμε να συζητήσουμε το εξάμεινο, το ευρωπαϊκό εξάμεινο. Σε αυτά τα πλαίσια κύριε Επίτροπε με τους συναδέλφους σας αποφασίσατε να καταστρώσετε τις κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση και ζητάτε την έγκριση του Κοινοβουλίου μας. Θέλουμε όμως να τονίσουμε τρία σημεία. Πρώτον, ως προς το περιεχόμενο της αιτήσιας αυτής έκθεσης για την ανάπτυξη. Μας εντυπωσιάζει το γεγονός ότι το θέμα της απασχόλησης και της ανεργίας φαίνεται σαν δευτερεύον σε σύγκριση με τους στόχους της δημοσιονομικής ενίσχυσης και για την αγορά της εργασίας έχουμε την εντύπωση ότι ζητάτε μια ρήξη του συμφώνου μεταξύ πολιτών και ένωση. Ζητάτε να αυξηθεί ο χρόνος εργασίας και να συνταξιοδότηση, να τροποποιηθούν οι συνθήκες εργασίας και να ανοίξουν ε, τα εμπορικά και τις Κυριακές. Νομίζουμε ότι όλα αυτά θα έχουν πολύ αρνητικές κοινωνικές επιπτώσεις και θεωρούμε επίσης ότι πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στους πιο ευάλωτους, τους νέους, τις γυναίκες, τους ηλικιωμένους ή τους αναπήρους. Επίσης θεωρούμε ότι υπάρχει μεγάλος κίνδυνος η δημοσιονομική αυτή γραμμή να αποτελέσει το α και το ω των στόχων σας. Δεύτερο σχόλιο. Με βάση αυτή την ετήσια εξέταση της ανάπτυξης, όπως είπατε και ο ίδιος, θα καθορίσετε εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων. Εκεί θα αποφασιστούν ακριβώς τα σημαντικά. Τι θα γίνει όμως για το ρόλο του Κοινοβουλίου σε όλα αυτά, ακόμη και αν εγκριθούν οι καινούργιες κατευθυντήριες γραμμές, πώς θα μπορέσει να υπάρξει μια δημοκρατική συζήτηση, πώς θα συνδυάσετε το 148 για το συντονισμό των προγραμμάτων απασχόληση με το 121 που μιλάει για συντονισμό της οικονομικής πολιτικής. Για μας υπάρχει μεγάλη σύγχυση εδώ διότι υπάρχει το θέμα της στρατηγικής του 2020 και οι εργασίες της ομάδας του κυρίου Βαν Ρόμπουη, η οικονομική δέσμη που συζήτησε ήδη το Κοινοβούλιο, τη μεταρρύθμιση, η αναθεώρηση της συνθήκης για τα δημοσιονομικά, αλλά επίσης και για μία πιθανή τους αλλαγή αρχίζεται το εξάμεινο αυτό τη στιγμή που η κυρία Μέρκελ και ο κύριος Σαρκοζή μιλούν για το σύμφωνο ανταγωνιστικότητας και άρα οι κατευθυντήρες αυτές γραμμές θα είναι κάτι το τελείως ασαφές. Επομένως κύριε Επίτροπε θέλω να σας επιστήσω την προσοχή στο τρίτο μας σχόλιο. Πέρυσι με συνενοχή της Βελγικής Προεδρίας καταφέραμε να κάμψουμε κάπως τις κατευθυντήρες γραμμές για την απασχόληση, ιδιαίτερα ως προς την διακυβέρνηση. Τι θα πει η διακυβέρνηση. Θα πει ότι δεν μπορεί να εφαρμοστεί οικονομική, κοινωνική, πολιτική επιτυχής αν δεν συνοδεύεται από πραγματική δημοκρατική συνεννόηση η οποία προϋποθέτει εξουσίες για το Ευρωπαϊκό και τα Εθνικά Κοινοβούλια και πραγματικό σεβασμό και συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους. Έχουμε την εντύπωση πολλές φορές ότι οι προτάσεις σας γυρίζουν την πλάτη σε όλα αυτά που είναι τα ουσιώδη στοιχεία της δημοκρατικής ζωής. Χωρίς συνειδητοποίηση των στοιχείων αυτών νομίζουμε ότι υπάρχει ο κίνδυνος να λείψει η συνοχή και οι λαοί μας να πάψουν να ενδιαφέρονται για αυτά που προσπαθούμε να πετύχουμε όλοι μαζί και να αποτύχει το κλειδί, δηλαδή το κοινοτικό πνεύμα, το ενωσιακό πνεύμα. Ευχαριστώ. Η κυρία Μπόουλς από την Οικονομική Επιτροπή. Πρόεδρος. Ευχαριστώ. Μπαίνουμε σε μια νέα εποχή οικονομικής διακυβέρνησης και η δομή του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου διαμορφώνεται αποτελώντας ένα από τα βασικά εργαλεία των καθηγητήριων γραμμών που προβλέπονται το, εφόσον συμπεριληφθούν τα 129 και 128 της συνθήκης στο κείμενό τους. Μέσα στο εξάμεινο η παρακολούθηση των, ε, μακρο, της μακροοικονομικής επιτυχίας και, των δημοσιονομικών προοπτικών μπορεί να συνδυαστεί με την στρατηγική Ευρώπη 20. Αυτό σημαίνει ότι το εξάμεινο μπορεί να παράσχει ένα συνεκτικό πλαίσιο για πολλές διαδικασίες οικονομικής διακυβέρνησης στην Ένωση, ενθαρρύνοντας ε, και τις δύο πλευρές. Ε, εκτενέστερα, η Οικονομική Υποτροπή υπογραμμίζει ότι η οικονομική διακυβέρνηση πρέπει να βασίζεται στην κοινωτική μέθοδο. Οι διαδικασίε θα πρέπει να είναι ανοιχτέ και να παρέχουν λογοδοσία αν θέλουν να έχουν την υποστήριξη των πολιτών. Τούτο απαιτεί την εμπλοκή και του Κοινοβουλίου όπου έπαιξε ρόλο το κοινοβούλιο, όπου παίζει ρόλο το κοινοβούλιο, πρέπει να έχει χρόνο να πληρεί την ε, δημοκρατική εντολή του. Η θέση της η ε, Οικονομικής Επιτροπής υποστηρίζει την ε, Επιτροπή Κοινωνικών Μημοθέσεων στο αίτημα αυτό. Για το ΕΛΚ, η κυρία Βότμαν Κόλ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε η χρηματοοικονομική κρίση κατέστησε σαφές ε, ότι η ανταγωνιστικότητά μας και έτσι και η κοινωνική οικονομία της αγοράς απειλούνται και γι' αυτό αυτό πρέπει να μάθουμε από την κρίση. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα την ενιαία εσωτερική αγορά μας. Πρέπει να διασφαλίσουμε το ότι θα λειτουργεί καλύτερα η αγορά εργασίας και γι' αυτό χαιρετίζει η ομάδα μου την Annual Growth Survey την ετήσια οικονομική ανάπτυξη στην αναθεώρηση και τα συμπεράσματα με ιδιαίτερα φιλόδοξο τρόπο σε σχέση με το εξάμεινο το οποίο έχουμε ενώπιόν μας. Σε σχέση με τις προσπάθειες αυτές είναι σαφές ότι χρειαζόμαστε μια Ευρώπη με αηφορία και ανάπτυξη, με επαρκή δημιουργία θέσεων απασχόλησης για τους πολίτες. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο με σταθερό νόμισμα και σταθεροποιημένη οικονομία, υπό τον όρο και προϋπόθεση ότι θα εξηγιάνουν τα οικονομικά τους, τα δημοσιονομικά τους, στα κράτη-μέλη διότι βλέπουμε ότι έχουμε προβλήματα αυτή τη στιγμή στα κράτη-μέλη με υπερχρέωση και υπερβολικά ελλείμματα και θα πρέπει έτσι να τεθούν τα θεμέλια για την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης ε, για, για την ανάπτυξη τα παιδιά μας και τις επόμενες γενναίες ε, που θα ακολουθήσουν. Κύριε Πρόεδρε, η ομάδα του ΕΛΚ εξακολουθεί να είναι πάντα υπέρ του πακέτου μέτρων για την οικονομική διακυβέρνηση με τρει άξονες. Ε, ένα σταθερό πλαίσιο συμφώνου σταθερότητας ε, με ε, επαρκή εποπτεία και αηφορία. Αυτό θέτει ως προϋπόθεση ότι θα υιοθετηθεί η κοινοτικοποιημένη μέθοδος ε, με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια. Αν επιτευχθεί αυτό δεν θα χρειάζεται πακέτο πλέον για την ανταγωνιστικότητα γιατί θα υπάρχει ήδη πλέον. Στη συνέχεια εξ ονόματος των Σοσιαλιστών ο κ. Ούντο Μπούλμαν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, εκπρόσωπε του Συμβουλίου, αγαπητοί ε, συνάδελφοι, άκουσα πολύ προσεκτικά διάβασα την έκθεση για την ανάπτυξη, διάβασα τα συμπεράσματα του Συμβουλίου ΕΚΟΦΗΝ και έχω συνειδητοποιήσει απόλυτα το εξή πλέον. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν βρίσκεται μόνο σε μια οικονομική κρίση, αλλά βρίσκεται σε μια πολιτική κρίση. Αυτά τα οποία μας συνιστάτε δεν είναι τίποτα το καινούριο από τους συνεργάτες σας ε, ζητήστε να σας υποβληθούν τα έγγραφα των τελευταίων δέκα ετών. Πάντα τα ίδια στοιχεία εμπεριέχονται. Πάντα τα ίδια αναφέρονται. Ότι είναι υπερβολικές λέει κρατικές δαπάνες. Πάντα όμω ε, αναφέρεται και ότι ο μηχανισμό ε, προσαρμογή θα πρέπει να στοχεύει στου μισθού που είναι, λέει, υπερβολικά υψηλοί. Δεν είδα άλλε συστάσει. Ό,τι, ό,τι και να συμβαίνει πάντα το ίδιο είναι ως σύσταση να μειωθούν οι μισθοί. Αυτό όμως δεν συσχετίζεται καθόλου με την πραγματική οικονομική κατάσταση των πραγμάτων. Σας υποβάλλω μια πρόταση. Στείλτε εκείνου που σα σημειώνουν όλα αυτά τα πράγματα, που κάνουν τι οικονομικέ αναλύσει στο Συμβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην Οικονομική και Νομισματική Κοινοβουλευτική Επιτροπή του δικού μα σώματο. Θέλουμε να συζητήσουμε μαζί σα για αυτά τα πρότυπα. Θέλουμε να δείτε αν βρίσκεται στα όρια τη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αν δείτε τα ποσοστά ανάπτυξη, θα κατανοήσετε για ποιο πράγμα κάνω λόγο. Και σα ερωτώ, γιατί δεν αναφέρετε τίποτα για τι επενδύσει με το χαμηλότερο ποσοστό επενδύσεων, το οποίο πλέον δεν είναι αηφόρο, όπου δεν υπάρχει καμία λέξη για τη βελτίωση των εσόδων ή για την ορθή ε, δίκαιη αντιμετώπιση της ε, κυκλικής αυτής ε, διαμόρφωσης των πραγμάτων. Ούτε λέξη δεν αναφέρεται για όλα αυτά. Έχετε χάσει τις ευκαιρίες και πρέπει να καταβάλλετε τεράστιες προσπάθειες να αρθείτε στο ύψος των προσδοκιών των πολιτών στην Ευρώπη. Σας λέω ένα πράγμα όμως. Αν αυτό είναι το πνεύμα με το οποίο εσείς θα λάβετε αποφάσεις το Μάρτιο, για την οικονομική διακυβέρνηση και το πακέτο μέτρων για τη μεταρρύθμιση του Συμφώνου Σταθερότητα δεν θα έχετε την ομάδα μα στο πλευρό σα ω σύμμαχο. Ευχαριστώ. Η κυρία Εκ για του φιλελεύθερου. Εκτός μικροφώνου. Σας ευχαριστώ. Πριν από ένα χρόνο εδώ μέσα μιλήσαμε για το τι έπρεπε να γίνει για να αντιμετωπίσουμε την σφαιρική συνολική χρηματοπιστωτική κρίση και είχαμε μιλήσει και για την οικονομική διακυβέρνηση. Σήμερα βλέπω με χαρά ότι πολλές από τις τοτινές μας συστάσεις έχουν πραγματοποιηθεί. Υπάρχει όμως ακόμη μεγάλο χάσμα μεταξύ των προσδοκιών και ευχών και των οικονομικών πόρων που διατίθενται για να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί στον προϋπολογισμό του προγράμματος 2020 πρέπει να μας εξηγήσει η Κομισιό, να μας ταυτίσει σαφώς ποιες δαπάνες θα χορηγηθούν για την επίτευξη της στρατηγικής αυτής. Αυτό ισχύει και για την επικείμενη αναθεώρηση του πολιετούς προγράμματος. Επίσης θέλω να απευθυνθώ κατευθείαν στα κράτη-μέλη. Δεν υπάρχει μεγάλη θέληση στο Συμβούλιο μεταξύ Υπουργών Οικονομικών και της δικής μου χώρας να επενδύσουν στο μέλλον οι εθνικοί προϋπολογισμοί πρέπει να δείχνουν ποιες είναι οι προσδοκίες του Συμβουλίου. Αλλιώς δεν πρόκειται ποτέ να επιτευχθεί τίποτα. Αν δεν έχουμε τα χρήματα εκεί όπου χρειάζονται δεν θα υπάρξει ανάπτυξη ούτε απασχόληση. Γι' αυτό ζητώ από την Κομισιόν να υποβάλει περισσότερες νομοθετικές προτάσεις και από τα κράτη-μέλη να δείξουν περισσότερη θέληση. Αλλιώς δεν πρόκειται να μεταφραστούν όλα αυτά στην πραγματικότητα σε τόσο σοβαρούς τομείς όπως την ενεργειακή αποδοτικότητα σε πανενωσιακό επίπεδο. Οι υπάρχουσες πρωτοβουλίες όπως το στρατηγικό σχέδιο για την ενέργεια, το σχέδιο μεγαλύτερης αποδοτικότητας έχουν εγκριθεί. Αλλά εσείς στο Συμβούλιο δεν φέρνετε τα χρήματα. Πώς θα χρηματοδοτηθούν αυτά τα προγράμματα. Όλοι συμφωνούμε να υπάρξουν περισσότερες θέσεις απασχόλησης και ανάπτυξη. Εμείς λοιπόν ως ομάδα ζητούμε από το Συμβούλιο, ε, δηλώνουμε προς το Συμβούλιο ότι δεν επιδεικνύει την απαραίτητη θέληση, πρέπει να επιστρέψουμε στην κοινοτική μέθοδο. Χαιρετίζω το, η μεγάλη συνένεση που υπάρχει για όλα αυτά στο Κοινοβούλιο, το οποίο σας δηλώνει ότι χρειάζεται δράση. Ευχαριστούμε ο κύριος Φίλιπ Λόμπερ των Πρασίνων. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, Συμβούλιο συνάδελφοι, ξέρετε ότι οι πράσινοι υποστηρίζουν μια πιο ενοποιημένη Ευρώπη, αποφασιστικά για να εξασφαλιστεί μια βιώσιμη ανάπτυξη για τους πολίτες μας, αλλά και για να ε, μπορέσει η Ευρώπη να σημαίνει κάτι στον 21ο αιώνα. Η εμπιστοσύνη μας ωστόσο σήμερα επηρεάζεται σοβαρά από μία πράξη που λάβατε, την ετήσια εξέταση ανάπτυξης, διότι αυτό είναι μία ιδεολογική θέση που είναι άσχετη με, ε, το, με τα γεγονότα. Τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι περικόπτουμε τις δαπάνες. Δεν επιβλέπουμε, περικόπτουμε τις εθνικές δαπάνες. Κάνουμε μεταρρυθμίζεται λέγεται, αλλά εμείς λέμε κάνετε ευέλικτη την αγορά εργασίας. Ε, όχι flexicurity, μόνο flexibility. Επιπλέον, μέτρα για το χρηματοοικονομικό τομέα. Δείτε το αυτό. Δείχνει τα, τα δύο μέτρα και δύο σταθμά. Τι λέτε για τα μέτρα, γρήγορα τα μέτρα, ισχυρά μέτρα. Για το χρηματοοικονομικό τομέα τι λέτε, λέτε μελέτη, εξέταση αντικτύπου, προβληματισμός και μεταβατική περίοδος ιδίω. Για την εξυγέννηση του προπολογισμού λέτε τώρα, εδώ και τώρα, ενώ για τις τράπεζες το 2019. Το ίδιο, και αφορά, το ίδιο αφορά και την ε, βιώσιμη ανάπτυξη. Δεν χρειαζόσαστε για περικοπές ε, μεταβατική περίοδο. Είπατε, πού είναι η Ευρώπη του 2020 όλα αυτά. Η Ευρώπη του 2020, κύριε Επίτροπε, κύριοι του Συμβουλίου, δεν είναι εφικτή με τις συστάσεις που κάνετε στα πλαίσια της ετήσιας ε, εποπτείας. Πραγματικά μας κοϊδεύεται όταν φαντάζεστε ότι μπορούμε να κάνουμε μια επενδυτική πολιτική όπως αυτή που απαιτείται στην έρευνα, στη φτώχεια, στη μείωση της φτώχειας, στην καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος και την απασχόληση με τις πολιτικές που συστήνεται. Αυτό είναι ψεύδι, η συζήτηση αυτή είναι θέατρο και μόνο. Ευχαριστώ για τους συντηρητικούς και μεταρρυθμιστές ο κύριος Χάρμπορ. Πρόεδρε, η ομάδα μου υποστηρίζει το ψήφισμα. Δεν σύμφωνουμε με όλα το περιεχόμενό του, αλλά το κύριο στοιχείο και το υπογραμμίζω και στο Συμβούλιο και την Επιτροπή, Μα βρίσκουν σύμφωνοι και συμφωνώ με τους τίτλους. Μία θαραλέα πράξη, ένας θηρίο νόμος ενίας πράξης και ένα νόμο για τι μικρέ επιχειρήσει για τη δημιουργία θέσεων εργασία. Από πού θα έρθουν οι δουλειέ, συνάδελφοι, από τι ιδιωτικέ επενδύσει, από τι ιδιωτικέ επιχειρήσει, από τι νέε εταιρείε. Ξέρουμε ότι οι μικρέ επιχειρήσει ήταν το βασικό εργαλείο δημιουργία θέσεων εργασία την τελευταία δεκαετία. Το μήνυμά μου προ όλου σα σήμερα είναι και τα 27 κράτη-μέλη πρέπει να ξεκινήσουν να θεωρούν σημαντικό το ζήτημα της δημιουργίας θέσεων εργασίας από τις επιχειρήσεις στο πλαίσιο της ενιαίας αγοράς. Έχουμε μια αγορά, τα κράτη έχουν επενδύσει για το άνοιγμα της, υπηρε... της αγοράς των υπηρεσιών, αλλά προώθησαν την, την ενιαία αγορά στις επιχειρήσεις, ενθάρρυναν τις επιχειρήσεις ε, ή το, online, το εμπόριο online. Γιατί δεν επιβάλλεται στα κράτη να κάνουν αυτά τα πρακτικά πράγματα για να απελευθερώσουν αυτά που υπάρχουν ήδη πέραν όλων των άλλων έργων που ανέφεραν οι συνάδελφοι. Σήμερα πρέπει να ξεκινήσει αυτό. Όχι να μιλάμε για κάτι άλλο που θα γίνει στο μέλλον. Ξεκινήστε να κάνετε δουλειά. Ο κύριος Μπίσκι. Ο πρόεδρος της Ενωτικής Αριστεράς. Κύριε Πρόεδρε, η συνάδελφος Χάμς χθε έθιξε ένα πολύ σημαντικό θέμα Κανένας δεν κατανοεί από τους πολίτες μας πια ποια στρατηγική, ποιοι μηχανισμοί σταθερότητας, ποιο σύμφωνο με ποιους και με ποιους κανονισμούς προτείνονται και θα τροποποιηθούν ή θα αρχίσουν να ισχύουν. Είναι σαφές ότι η στρατηγική για την Ευρώπη του 2020 δεν έδωσε λύσεις για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες μας μέσα σε αυτή την κρίση. Το αντίθετο, συνεχίζονται οι λαθασμένες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συνεισέφεραν σε αυτή την κρίση. Συνεχίζουν να στοιχηματίζουν υπέρ του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Θα γίνει, λέει, πιο αυστηρό αυτό το πλαίσιο με μηχανισμούς κύρωσης Ουσιαστικά πρόκειται για πολιτικές εξοικονόμησης κονδυλίων εις βάρος των πολιτών, πολιτικές λιτότητας, παράταση του χρόνου εργασίας. Είτε τώρα αυτό σε σχέση με τους μισθούς, είτε με τις διαπραγματεύσεις με τους κοινωνικούς εταίρους θα οδηγήσουν σε κάποιους περιορισμούς ή στην ελαστικοποίηση του χρόνου εργασίας, θα πρόκειται για μισθολογικές περικοπές και περικοπές γενικά. Και πρόκειται και για παρεμβάσεις στην οικονομική δραστηριότητα της κοινωνίας. Κάποιοι κάνουν λόγο για το χειρόφρενο έναντι της υπερχρέωσης. Είναι αδιάφορο αν αυτό το αποκαλεί κανείς οικονομική διακυβέρνηση οικονομική διακυβέρνηση ή σύμφωνο πολιτικής σταθερότητας και ανάπτυξης ή σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με βάση την ετήσια οικονομική ανάπτυξη. Αυτές οι κατά της κοινωνικής πολιτικής πολιτικές δεν τις υποστηρίζει η ομάδα μου αλλά διαφοροποιείται η υπόθεση αν το κοινοβούλιο και τα κοινοβούλια έχουν κάποιο λόγο να αρθρώσουν σε αυτό το πλαίσιο ή όχι σε σχέση με τις δυνατότητες ε, οι ευρωβουλευτές ε, να μπορέσουν να υποβάλουν μια πρόταση ώστε σε σχέση με την ενκρυπτό και παραβίστο πολιτική των κυβερνήσεων όπως ακολουθεί το να μπορέσουμε να παρέμβουμε εμείς και δεν θα έπρεπε να δεχθούμε μια οπισθοχώρηση, οπισθοδρόμηση σε μια Ευρώπη δύο ταχυτήτων. Ευχαριστώ. Thank you. Ε, Mr. Mario... κύριος Μποργέζιο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Η Ευρώπη 2020 είναι τεράστιο πρόγραμμα αλλά Είμαστε βέβαιοι ότι θα πετύχουμε το στόχο μας τότε. 20% ανανεώσιμη ενέργεια. Αμφίβολο είναι και λόγω της κρίσης που ε, επιβραδύνει τις επενδύσεις. Επιπλέον υπάρχει το πρόβλημα ε, των επιδοτήσεων στην Κίνα που είναι η πρώτη εξαγωγός χώρα των φωτοβολταϊκών πάνελ. Θα έπρεπε να ενθαρρύνουμε, αυτό πρέπει να κάνουμε, την έρευνα και την παραγωγή φωτοβολταϊκών πάνελ στην Ευρώπη, ιδίως δημιουργώντας οικονομίες κλίμακος υιοθετώντα μαζικά φερρυπίν τέτοια πάνελ στι ε, πόλει τη Ευρώπη. Κάτι διαφορετικό θα έπρεπε να κάνουμε, να δημιουργήσουμε μια ευρωπαϊκή, πανευρωπαϊκή εταιρεία ε, ηλεκτρισμού υπομορφήν δημόσια ε, εταιρεία. Ε, δεδομένου ότι τα δίκτυα διανομής και οι υποδομές τους σήμερα αποτελούν υφιστάμενα φυσικά νομοπόλια, θα έπρεπε να έχουν ενιαία διαχείριση. Αντίθετα, προτιμήσαμε να δώσουμε λόγω μια υπερβολικού φιλελευθερισμού ε, ε, διαφορετικές λύσεις που δεν είναι προς όφελος των καταναλωτών αλλά των μετόχων των μονοπωλίων. Εδώ και 150 χρόνια δεν μειώνεται η παραγωγή του διοξιδίου του άνθρακα στην Ένωση, διακόπτει τον συνεχίζω μιλητής. Έρευνα για οχήματα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κλέης. 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. για να μπορέσουμε να πετύχουμε τους στόχους απασχόλησης για τη στρατηγική Ευρώπη 2020. Είναι σημαντικό η πολιτική για τη μετανάστευση των περισσότερων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ρυθμιστεί σωστά. Το ανέφερε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι προτεραιότητες είναι ενισχυμένο ποσοστό απασχόλησης, μείωση της διαθροτικής ανεργίας, ανάπτυξη των καταρτισμένων εργαζομένων που θα μπορέσουν να δραστηριοποιηθούν στην αγορά εργασίας, διαβίω εκπαίδευση και μάθηση, εισαγωγή μαζικά ε, χειρών εργασίας ε, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Ευρωπαϊκή Ένωση δείχνει μια κοντόθωρη αντιμετώπιση και είναι το αντίθετο της προσέγγισης που ανέφερα. Υπάρχουν 25 εκατομμύρια άνεργοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να ξεκινήσουμε αυτού του ανθρώπους να τους οδηγούμε στην απασχόληση αντί μαζικά να ευνοούμε την μαζική μετανάστευση. Και έτσι τώρα το να φέρουμε κατατισμένους εργαζόμενους στην Ευρώπη, το brain drain αυτό, η αποστράγγιση εγκεφάλων δημιουργεί προβλήματα σε σχέση με ε, χώρες και που θα παραμένουν σε μάσα εργαζόμενοι οι οποίοι δεν θα έχουν κατατιστεί σωστά. Χρειάζεται μια ανάλυση κόστους-οφέλους όσον αφορά την μετανάστευση από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτή η πτυχή θα πρέπει να αποτελέσει μέρος των κατευθυντήριων γραμμών για την απασχόληση. Ευχαριστώ. Άλλοι ομιλητές. Ο κύριος Μαρινέσκου, 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Η στρατηγική του 2020 περιλαμβάνει στόχους που δεν μπορούν να επιτευχθούν εάν δεν δοθεί η απαραίτητη σπουδότητα σε κάποιες διαστάσεις, σε κάποιε πτυχέ πτυχές Τη γεωργία για παράδειγμα, με τη συμβολή του, στη βιώσιμη ανάπτυξη και τη συμπερίληψη τη γεωργία στον τομέα αυτό, καθώς και την ανάγκη ε, ε, αξιόπιστης παραγωγής ε, ειδών διατροφής, διαφύλαξης των εδαφικών, της εδαφικής διαφορετικότητας και της ανάπτυξης πέθου. Όλα αυτά είναι αναγκαία για έναν παραγωγικό αγροτικό τομέα. Σε ό,τι αφορά τη βιομηχανική πολιτική, υποδομέ υποδομές, η δημιουργία ενός ενιαίου σιδεδομικού χώρου είναι αναγκαίο για την ε, αύξηση των σιδεδομικών μεταφορών. Επιπλέον θα πρέπει να ολοκληρωθεί ο, το, ε, ο ενιαίος ευρωπαϊκός ουρανός και το ε, πρόγραμμα Γαλιλαίο. Επίσης να αυξηθούν οι, τα ευρωπαϊκά δίκτυα, όχι μόνο στις μεταφορές αλλά και στα ενεργειακά δίκτυα με την με τους απαραίτητους πόρους τα έργα αυτά που έχουν προστιθέμενη ευρωπαϊκή αξία. Για παραδείγμα, το Ναμπούκο, το οποίο θα έχει πλονεκτήματα για όλα τα κράτη-μέλη, μειώνοντας την εξάρτηση της Ένωσης από πηγές ενέργειας εκτός Ένωσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Συνεχίζουμε τον κατάλογο των ομιλητών. Το λόγο θα πάρει η κυρία Ουρσκοτ για 1,5 λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αν θέλουμε μετά την κρίση να αναθερμαθεί η οικονομία πρέπει να δημιουργηθεί αξιοπιστία. Ο Ριχάρδος Βίλκινσον, ένας Βρετανός ερευνητής που έχει γράψει πολλά άρθρα και ήρθε να μας μιλήσει την περασμένη εβδομάδα στις Βρυξέλλες, μας είπε ότι χρειάζεται μεγαλύτερη ισότητα για να μπορέσει να υπάρξει αξιοπιστία. Η στρατηγική του 2020 πρέπει να δημιουργήσει την αξιοπιστία αυτή. Αν θέλουμε να πετύχουμε το στόχο αυτό πρέπει να συμμετάσχουν και τα συνδικάτα. Η κρίση αφορά τους εργαζόμενους και τα συνδικάτα και τους συνταξιούχους. Εμείς οι γυναίκες στην Ευρώπη πρέπει να έχουμε τις ίδιες δυνατότητες με τους άντρες. Αυτό δεν το λέει πάντα ρητά το ψήφισμα. Πρέπει όμως να εφαρμοστεί, να πραγματοποιηθεί. Τρίτον, πρέπει να ενδυναμωθεί βιομηχανική πολιτική και να υπάρξουν επενδύσεις στο μέλλον, στις υποδομές. Να υπάρξει δηλαδή πολύ καλύτερη χρήση των πόρων που διαθέτουμε για να δημιουργηθούν περισσότερες πράσινες θέσεις απασχόλησης ή θέσεις πράσινης απασχόλησης. Τέταρτον, πρέπει να γίνει μια μεγάλη προσπάθεια εξοικονόμησης ή μεγαλύτερης αποδοτικότητας στην ενέργεια. Σήμερα οι στόχοι που έχουμε θέσει δεν είναι δεσμευτικοί, πρέπει όμως να γίνουν. Είναι κάτι ουσιώδες αν θέλουμε να πετύχουμε το στόχο της μεγαλύτερης ανταγωνιστικότητας που είναι ο κόμβος της στρατηγικής 2020 αν δεν επιδείξουμε τέτοια φιλοδοξία δεν θα υπάρχει και πολιτική θέληση. Ιδιαίτερα στον τομέα της ενέργειας όπου πρέπει να γίνει εξυπνότερη χρήση των πόρων για να πληρώνουν λιγότερα οι καταναλωτές και καταναλώτριες και ταυτόχρονα να ενδυναμώνεται η δραστηριότητα των επιχειρήσεων. Η κυρία Λίνε για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ. Αν θέλουμε την στρατηγική Ευρώπη 2020 να πετύχει, τότε οι καθηγητές γραμμές πρέπει να υλοποιηθούν αποτελεσματικά και τα εθνικά μεταρρυθμιστικά προγράμματα να ε, τεθούν σε ισχύ και να λάβουν την προτεραιότητα που τους αρμόζει. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι κανείς δεν μένει πίσω. Η ανεργία μεταξύ των ατόμων με αναπηρίες ή των ηλικιωμένων είναι ε, επονίδιστες και τα κείμενα αναφέρονται στην ανάγκη να υλοποιηθούν στο χώρο εργασίας η νομοθεσία κατά, της, κατά των διακρίσεων. Είναι σημαντικό οι στόχοι που συμφωνήθηκαν σε ευρωπαϊκό επίπεδο να υλοποιηθούν. Και βεβαίω τα κράτη-μέλη είναι αυτά που θα θέσουν συγκεκριμένου στόχου και θα του στηρίσουν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, ωστόσο, παίζει σημαντικό ρόλο για την βελτίωση των ανταλλαγών βέλτιστων πρακτικών. Και γι' αυτό η παράγραφο 27 του ψηφίσματο τη Επιτροπή είναι σημαντική και το καθιστά σαφέ έχουμε μήνες εσωτερικών συζητήσεων για το, τη μορφή της στρατηγικής Ευρώπης 2020. Έχουμε ωστόσο τι οδηγίε, τι καθηληφτήρες γραμμέ για την απασχόληση. Ας αρχίσουμε να τις υλοποιούμε. Ευχαριστώ πολύ κυρία Λίνε. Τώρα το λόγο θα πάρει η κυρία Τούρουνεν για 1,5 λεπτό παρακαλώ. Øh, Σας ευχαριστώ πολύ. Πολλής λόγος γίνεται εδώ για την ευθύνη στα οικονομικά θέματα και την υπευθυνότητα μέσα σε αυτή την οικονομική συγκυρία στην Ευρώπη. Πολύ συχνά όμως αυτό είναι μια παρέμβαση για τις δημόσιες δαπάνες και πολύ σπάνια συνδέεται αυτό με βελτίωση στην κατάσταση απασχόλησης. Πρέπει να ρωτήσουμε τι είναι λοιπόν η οικονομική υπευθυνότητα. Εμείς οι πράσινοι βλέπουμε τεράστια αντίφαση όσον αφορά τις πολιτικές που ακολουθούνται στην Ευρώπη και στα κράτη-μέλη. Αφενός το βλέπουμε στην ετήσια έκθεση για την ανάπτυξη και για το οικονομικό εξάμεινο, για την ευρωπαϊκό εξάμεινο. Και όλο και λιγότερη ανάπτυξη σημειώνεται και λιγότερε θέσει απασχόληση επιτυγχάνονται. Από την άλλη πλευρά, λέμε ότι έχουμε την στρατηγική για την Ευρώπη του 2020 και τι κατευθυντήριε γραμμέ για την δημιουργία περισσότερων θέσεων απασχόληση και ανάπτυξη. Αυτά όλα δεν αντιστοιχούν το ένα προ το άλλο. Έχουμε εκατομμύρια ανέργους στην Ευρώπη μεγάλος τεράστιος αριθμός είναι νέοι άνθρωποι. Είναι φτωχοί άνθρωποι που υπάρχουν στην Ευρώπη και δεν βελτιώνεται η κατάσταση οικονομικά με όλα τα μέτρα που λαμβάνονται. Το αποφασιστικό είναι εδώ να δημιουργηθούν νέες θέσεις απασχόλησης στην Ευρώπη και πραγματικά να υλοποιηθούν οι στρατηγικές για την Ευρώπη του 2020 και για την πολιτική για την ανάπτυξη και να γίνουν όλα αυτά στην οικονομική πολιτική χειροπιαστά. Αυτό θα ήταν κάτι θετικό, αλλά φοβούμαι δεν θα επιτευχθεί. Κύριος Καμπρονόχο, αλλά δεν φαίνεται στην αίθουσα και θα πάρει το λόγο ο κύριος Αλαβράκος για ένα λεπτό. Πρόεδρε, η φτώχεια, οι κλιματικές αλλαγές, η υπογεννητικότητα, η μετανάστευση, η ενέργεια, αλλά κυρίως η αντιμετώπιση της ανεργίας είναι τα προβλήματα που έχουμε σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση η αντιμετώπιση τους χρειάζεται χρήματα χρειάζεται πιστώσει, σε όλη όμω την ευρώπη δυστυχώς παρουσιάζεται πιστωτική συρρήκνωση. τι σημαίνει αυτό; η στρατηγική 2020 είναι επισφαλής είναι δύσκολο να επιτύχει. πρέπει όμως να προσπαθήσουμε. θεωρώ ότι ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δώσουμε στην ανεργία τα ποσοστά τη οποία είναι τα μεγαλύτερα τη τελευταία δεκαετία. θεωρώ επίση ότι πρέπει να δώσουμε ποιοτική εκπαίδευση στου νέου τη Ευρώπη που να εναρμονίζεται στι ανάγκε τη εργασία και τα εκπαιδευτικά προγράμματα πρέπει να μεταρρυθμιστούν ει τρόπον ώστε τα κράτη μέλη να δεσμευτούν για τη μείωση τη πρόορη εγκατάλειψη των σπουδών. οι κενέ θέσει εργασία απαιτούν εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό. καλώ την ευρώπη να θεσπίσει χωρί καθυστέρηση το προτινόμενο ευρωπαϊκό σύστημα παρακολούθηση κενών θέσεων που να περιλαμβάνει επίσης ένα ευρωπαϊκό διαβατήριο δεξιοτήτων. πρέπει να επιτύχουμε. οι λόγοι δεν αρκούν πρέπει να κάνουμε πράξεις. ευχαριστώ κύριε πρόεδρε. Λόγο τώρα για λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Υπάρχει μία ερώτηση, μία και μόνη ερώτηση τι μπορούμε να κάνουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο προκειμένου να έχουν εργασία αυτοί που δεν έχουν αυτή τη στιγμή. Για να απαντήσουμε σε αυτή την ερώτηση θα πρέπει να υπάρχει σαφή συνένεση στο γεγονός ότι δεν υπάρχει ανάπτυξη χωρίς μακροοικονομική σταθερότητα. Κάποια από τα πράγματα τα οποία προτάθηκαν κυρίως ε, από την αριστερά θα ήταν ψωμίχια σήμερα και πείνα για το αύριο. Δεύτερον, η Ευρώπη του 2020 είναι ένας κατάλογος καλών προσθέσεων, ωραία μουσική, αλλά πρέπει από τις μουσες να περάσουμε στο θέατρο. Τι θα κάνουμε και πώς θα χρηματοδοτήσουμε τις ε, πρωτοβουλίες και τις δράσεις που προτείνονται εδώ συνάδει η φιλοδοξία της στρατηγικής του 2020 με τους περιορισμούς που μας ανακοινώνονται στον προϋπολογισμό. Και τρίτο στοιχείο, για να μπορέσουμε να έχουμε σταθερή ανάπτυξη θα πρέπει να υπάρχει σαφής εικόνα. Και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει πλήρης εικόνα. Αυτά τα οποία γίνονται στο ΕΚΟΦΗΝ ε, τις τελευταίες ημέρες είναι διαπίστωση ότι έχουμε διάσπαρτες ιδέες εδώ και εκεί, ε, αλλά δεν υπάρχει σαφήνεια. Υπάρχουν τρία σημαντικά πράγματα. Δεν θα πρέπει να ε, αφήσουμε καταρχά τι χώρε οι οποίε διαπιστώνουν δυσκολίε αυτή τη στιγμή. Θα πρέπει να υπάρχει συνεχή στήριξη. Επίση, θα πρέπει να προχωρήσουν ε, τα συγκεκριμένα στοιχεία που προτείνονται στην έκθεση Μόντι, αλλά δεν παρουσιάζονται στη στρατηγική του 2020. Και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, που έχει πόρου στα δύο τρίτα του πόρου Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα πρέπει να προχωρήσουν και θα έχουν τα ίδια χρήματα που είχαν στο σχέδιο ε, Marshall για την της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ξεφεύγει κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Η κυρία Ποδηματά τώρα για 1,5 λεπτό παρακαλώ κύριε πρόεδρε εδώ και μήνες συζητάμε στην ένωση για μια αποτελεσματική συνεκτική και βιώσιμη απάντηση στην κρίση μια απάντηση που θα διασφαλίσει την επίτευξη των στρατηγικών μας στόχων που είναι η βιώσιμη ανάπτυξη η προστασία της απασχόλησης η κοινωνική πρόοδος και η κοινωνική συνοχή. υπάρχουν όμως δύο προβλήματα. πρώτον η συζήτηση για τη στρατηγική 2020 εξακολουθεί να είναι οργανικά ξεκομμένη από το πακέτο της οικονομικής διακυβέρνησης από το ευρωπαϊκό εξάμεινο από την ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης με αποτέλεσμα να έχουμε είτε μια κατακαιρματισμένη στρατηγική είτε παράλληλες στρατηγικές στρατηγικές που τρέχουν παράλληλα χωρίς επαρκή συντονισμό με αποτέλεσμα και κίνδυνο να υπονομεύει μία την άλλη το δεύτερο πρόβλημα είναι ότι η έμφαση σήμερα από την πλευρά του συμβουλίου και της ευρωπαϊκής επιτροπής είναι στην αυστηροποίηση των κανόνων του συμφώνου σταθερότητας και ανάπτυξης και στην δημοσιονομική πειθαρχία και προσαρμογή χωρίς να υπάρχουν πιστικές απαντήσεις και λύσεις για την αποτελεσματική εφαρμογή και την χρηματοδότηση των στόχων της στρατηγικής. 2020 κυρίε και κύριοι συνάδελφοι πιστεύω ότι υπάρχει κίνδυνο όπω έγινε και με τη στρατηγική της Λισαβόνας, πολλοί από τους στόχους μας να μείνουν στα χαρτιά και και φοβούμαι ότι αυτό θα συμβεί εάν δεν είμαστε πιστικοί απέναντι στους ευρωπαίους πολίτες που σηκώνουν το βάρος της κρίσης που δεν μπορούν ούτε οφείλουν να παρακολουθήσουν τις τεχνικές συζητήσεις για τη μεταρρύθμιση του συμφώνου σταθερότητας για τους δείκτες και τις κυρώσεις. πρέπει να αντιληφθούμε ότι δεν μπορούμε να ασχολούμαστε μονομερώς με δείκτες και αριθμούς πρέπει να ασχοληθούμε με τους ανθρώπους. Ευχαριστώ το λόγο τώρα θα πάρει η κυρία, Γκουλάχ για ένα λεπτό. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, αν θέλετε, εκπρόσωπο τη ε, Προεδρία, μπορείτε να με ακούσετε. Κύριε Επιτρόπε, έχω ένα λεπτό και παρόλα αυτά θα ήθελα να σιωπήσω. Να μην πω τίποτα. Γιατί αυτή η στρατηγική του 2020 έχει απομακρυνθεί από αυτό που χρειαζόμαστε. Μας κοροϊδεύετε με τα λόγια. Πιστεύετε ότι μια κατευθύνια γραμμή με κάποια με κάποιες ιδέες που αναπτύσσετε και σας απασχολούν εδώ και πολλές μέρες, θα δώσουν εργασία στους Ευρωπαίους. Κάνετε λάθος. Για κοίταξε τι γίνεται στον κόσμο. Δεν νομίζω ότι οι Κινέζοι, οι Ινδοί ή οι αναπτυσσόμενες χώρες εντυπωσιάζονται αυτά που κάνουμε για την ανάπτυξη. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να σιωπήσω ενώπιον ημών και να σας πω ένα πράγμα. Θα είμαστε πολύ αυστηροί στην εργασία μας. Ας μην νομίζει το Συμβούλιο ότι αρχίζει να μας πει να επιταχύνουμε για να πιστεύω ότι θα έχουμε συμφωνία τον Ιούνιο. Θα έχουν συμφωνία όταν έχει ζητήσει το θέμα στο Κοινοβούλιο, όταν μας έχει ακούσει το Συμβούλιο και τα ευρωομόλογα θα μπορέσουν να δημιουργήσουν μια παγκόσμια αγορά και αυτό θα πρέπει να είναι τμήμα γι' αυτό της ελόγω Ευχαριστώ. Τώρα για ένα λεπτό ο κύριος Έπνικ θα πάρει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, νιώθω λίγο αμήχανα με την φρασιολογία που χρησιμοποιείται εδώ. Η οικονομική ανάπτυξη έχει κάποιες προϋποθέσεις και βλέπουμε ότι οι κυβερνήσεις δεν δημιουργούν θέσεις απασχόλησης. Υπάρχει έλλειμμα ανταγωνιστικότητας ε, και υπάρχει 35% διαφορά ως προς την ανάπτυξη ανάμεσα στον Βορρά και στον Νότο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, εντάξει το σύμφωνο ανταγωνιστικότητας, αλλά κοιτάξτε η συνθήκη της Λισαβόνας η στρατηγική της Λισαβόνας μάλλον, διορθώνει ο μιλητής, δεν έχει αποφέρει καρπούς. Δεν μπορούμε να επιβάλλουμε αυτά τα πράγματα στις ε, κοινωνίες στην κοινωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, θα καταστρέψουμε τις θέσεις απασχόλησης ε, που υπολείπονται σε 21 χώρες βάσει δημοσκοπήσεων υπάρχει ένα ρεύμα κατά της φορολόγησης των επιχειρήσεων. Δεν ο τώρα Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε, συνάδελφοι, βρισκόμαστε μέσα σε μια μεγάλη οικονομική κρίση. Ζητάμε το κείμενο, σωστό είναι. Αλλά συνήθω συζητάμε με τίτλου και μετά κλείνουμε το στόμα, σαν να μην έχει γίνει τίποτα. Αυτό οφείλεται στο γεγονό, νομίζω, ότι εδώ στο Κοινοβούλιο εμεί δεν είμαστε αρκετά ειλικρινεί ακριβώς κάνουμε μία πολιτική τίτλων. Γιατί πρέπει να αναπτύσσουμε την ε, ανάγαμψη, τη σταθερότητα. Ας κάνουμε κάτι συγκεκριμένο. Ας εξετάσουμε κριτικά κατά πόσον δαπανούμε τα χρήματά μας σωστά. Ή κάθε μέρα ο καθένας μας έχει μια καινούργια τίτλο. πώς θα μπορέσουμε να δαπανίσουμε χρήματα. Άμα μπορέσουμε τους σπόρους μας να τους συγκεντρώσουμε στα μελλοντικά προγράμματα, τότε μόνο θα καταφέρουμε να προχωρήσουμε. Γιατί δεν είναι σωστό να διαθέτουμε εδώ και εκεί κάποιους πόρους. Θα πρέπει να ακολουθήσουμε μια πολιτική που να ενθαρρύνει τη βιομηχανία και όχι να σκεφτόμαστε από το πρωί μέχρι το βράδυ πώς θα τους παρενοχλήσουμε. Από το πρωί μέχρι το βράδυ υιοθετούμε νέες αποφάσεις που παρεμποδίζει την εξέλιξη της οικονομίας. Ε, Παραδείγματο υπάρχει τίποτα για δεσμευτικά μέτρα για την αποτελεσματική ενέργεια Πιστεύετε ότι με τις αποφάσεις που περνάμε εδώ για την ενέργεια μπορέσουμε να προωθήσουμε την, την οικονομία ή την παρεμποδίζουμε. Και θα ήθελα να το σκεφτούμε το θέμα πιο ειλικρινά, να πάρουμε πιο λίγες αποφάσεις, αλλά εκείνες τις αποφάσεις που θα μας βοηθήσουν να προχωρήσουμε. Είναι πιο δύσκολο, πιο κοπιαστικό, θα τσακωθούμε, αλλά αυτή είναι η έννοια της δημοκρατίας. Κυρία έχει λόγο για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Η χρηματοοικονομική κρίση έχει γίνει πλέον μια κρίση απασχόλησης, κρίση της αγοράς εργασίας. Γι' αυτό και με χαροποιεί το γεγονός ότι στην Ευρώπη αντιληφθήκαμε ότι υπάρχει ανάγκη συντονισμού και σε θέματα πολιτικής απασχόλησης για την οικονομία. Αυτό σημαίνει ότι απαιτούνται φορολογικές μεταρρυθμίσεις, μεταρρυθμίσεις στην απασχόληση. Εάν μια χώρα λάβει μέτρα προς αυτό το τομέα, ε, ακόμα και αν τροποποιήσει το, η νομοθεσία για το άνοιγμα των καταστημάτων ε, και το ωράριο των καταστημάτων, θα πρέπει πάντα να έχει κατά νου και πώς θα επηρεάσει αυτό την απασχόληση. Κάθε απόφαση λοιπόν έχει τη σημασία της και αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι θα πρέπει να γίνεται και από κοινού με την ε, κοινή ε, συμφωνία και με τους κοινωνικούς εταίρους. Εκείνο επίσης που θα είναι σημαντικό είναι και η πρώτη στιγμή επαλήθευσης των ε, μέτρων ε, και αυτών των πρωτοβουλειών όταν ε, θα γίνει ένας απολογισμός της κατάστασης και θα εξεταστούν τα αποτελέσματα. Ελπίζουμε αυτό να γίνει στη διάρκεια της Ουγγρικής Προεδρίας και η Ουγγαρία λοιπόν έχει διτό ρόλο και ως Προεδρεύουσα αλλά και ως χώρα η οποία θα πρέπει να δίνει το παράδειγμα. Όταν λαμβάνονται αποφάσεις θα πρέπει να λαμβάνεται πάντα αυτό υπόψη. Λοιπόν, κυρίε και κύριοι συνάδελφοι, έχουν ζητήσει blue card, ε, δηλαδή το δικαίωμα που έχουν να παρέμβουν στην ε, συζήτηση. Καταρχά, ε, καταρχάς, η κυρία Μορβάη. έχετε το λόγο, κυρία Μορβάη, πολύ σύντομα σας παρακαλώ. Πρώτα ζήτησε η κυρία Μορβάη. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρία Κιόντς, φαίνεται ότι κατανοεί την, ε, τα προβλήματα και ξέρει πώς δημιουργούνται θέσεις απασχόλησης. Ίσως εγώ όμως κάτι να παρανόησα. Θα μπορέσετε λοιπόν να με βοηθήσετε. Από πού θα προέρθουν τα χρήματα αυτά, πού θα δημιουργηθούν αυτές οι θέσεις απασχόλησης, αυτές οι ερωτήσει για τις οποίες ευχαρίστω θα ήθελα μια απάντηση. Ίσως και ο Σύμβουλο να μπορεί να απαντήσει σε αυτά. Ή και ο κύριο Επίτροπο. Και αυτό ισχύει όχι μόνο για την Ουγγαρία αλλά και για άλλε ευρωπαϊκέ χώρε. Πώ μπορούμε πραγματικά να δημιουργήσουμε τι θέσει αυτέ τη απασχόληση. Και άλλη μια ερώτηση, από πού θα προέρθουν αυτές τις θέσεις απασχόλησης. Παρακαλώ συγκεκριμένη απάντηση. Επί να κρατήσουμε το περιεχόμενο του δικαιώματο με την μπλε κάρτα. Η, δεν, μπλε κάρτα δεν είναι μια ερώτηση γενικά που απευθύνεται στην ε, Ολομέλεια, στον Επίτροπο ή στον εκπρόσωπο του Συμβουλίου. Απευθύνεται σε έναν συνάδελφο που ε, ε, αναπτύσσει ένα θέμα για το οποίο θέλετε να ζητήσετε μια διευκρίνηση. Λοιπόν, κυρία Μορβάη, δεν ήταν αυτό το πνεύμα της ερώτησής σας. Ε, τώρα έχει ζητήσει... Α, η κυρία Γκόντς θέλει να απαντήσει σε αυτό το θέμα, μια και ενδιαφερθήκατε για αναφερθήκατε στην Ουγγαρία. Κυρία Γκόντς, θέλετε να δώσετε μια πολύ σύντομη απάντηση στην κυρία Μορβάη σε κάτι που έχει σχέση με την παρέμβαση που μόλις κάνατε. Ναι. Eh, Ευχαριστώ. Παρόλο που δεν έχω αρκετό χρόνο, δεν μπορώ να το αναπτύξω το θέμα αυτό στις λεπτομέρειες του, αλλά φαντάζομαι ότι όταν παραδείγματος θα αλλάξει κάτι με την, σχετικά με τη φορολογία. Αυτή είναι μια δημιουργία δημιουργία θέσεων απεσχόλησης. και η εξάλληψη των διαφορών ότι μπορούμε να βοηθήσουμε δηλαδή τις επιχειρήσεις, να του δώσουμε κάποια κίνητρα για να μπορέσουν να δημιουργήσουν αυτέ τι θέσει απασχόληση. Όλα αυτά θα μπορούσαν να προωθηθούν. Είναι δυνατόν νομίζω με αυτόν τον τρόπο να δημιουργηθούν θέσεις απασχόληση. Το ίδιο εάν τροποποιήσουμε το σύστημα τη παιδεία και τη εκπαίδευση. Και αυτό είναι μια δημιουργότητα και είναι σημαντικό και για την ολοκλήρωση, την εσωμάτωση όλων των πολιτών. Εκπαίδευση, παιδεία, μετεκπαίδευση και δεν αυτά ζητήσει να παρέμβει με blue card. Kiitoksia. Ε, kun kollega siellä oikealla väitti kiveen kovaan, että... Η συνάδελφός μου ισχυρίζεται ότι με την πολιτική αναταράσουμε την οικονομία. Μα το πιστεύει πραγματικά πραγματικά πιστεύει ότι ε, προσπαθώντας να οργανώσουμε την οικονομία το μόνο που κάνουμε είναι να την αναταράσουμε. Κύριε Ρόλ, θέλετε να απαντήσετε σύντομα, 30 δευτερόλεπτα. Μόνο σύντομα. Ναι. Εάν δείτε τα μέτρα που υιοθετήθηκαν τους τελευταίους μήνες, τα συναθρήσετε και δείτε πόσο κόστος δημιουργήσαμε έτσι, πολλές φορές αυτό οδήγησε στην διατάραξη της εξέλιξης της οικονομίας και αυτό θα πρέπει να το σκεφτούμε. Και γι' αυτό η συμβουλή του Επιτρόπου Βιομηχανίας ήταν πάρα πολύ ευφύς. Δηλαδή στις μελλοντικές αποφάσεις να κρίνουμε πώς αυτές θα έχουν επιπτώσεις στην ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα. Ο Πέζης του Ριτς White ζήτησε επίσης να παρέμβει ε, στον κύριο Ρόλ. Θέλετε το λόγο, κύριε Στουρίτς, θέλετε, εξακολουθείτε να θέλετε το λόγο. 30 δευτερόλεπτο, παρακαλώ. Δεν βλέπω να αντιδρά ο κύριο Ιστουρίτς. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ο κύριος Σίμπερ θα πάρει το λόγο τώρα για 1,5 λεπτό. Ε, Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Όλοι γνωρίζουν εδώ όσο πιο πολύ συνενώνεται η Ευρώπη, τόσο πιο πολύ θα υπάρχει συμφωνία στο οικονομικά θέματα. Και αυτό, αυτό το μέσο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου είναι λογικό, αλλά θα πρέπει να σταματεί εκεί που παρεμβαίνει σε θέματα που είναι αρμοδιότητα των κοινωνικών εταίρων παραδείγματο χάρη διαπραγματεύσει για τι μισθολογικέ εξελίξει. Εδώ θα πρέπει να απόσχουμε από την παρέμβαση, γιατί δεν είναι σωστό να κοιτάει η Ευρώπη που υπάρχουν οι πιο ψηλοί μισθοί και να του ακολουθεί αυτού. Θα πρέπει εδώ να εξαλείψουμε τα εμπόδια για να μπορέσει να ανθίσει η ευρωπαϊκή οικονομία. Αυτό αφορεί ολιγοπόλια και μονοπόλια, αλλά και παρεμποδίσει για την πρόσβαση στην αγορά. Δεν επιτρέπεται ορισμένε ορισμένοι κλάδοι να έχουν εξασφαλισμένα περιθώρια κέρδους. Θα πρέπει να δώσουμε δυνατότητα στην ευρωπαϊκή οικονομία να αναπτυχθεί ξεκάθαρα. Θα πρέπει επίσης να καινοτομήσουμε όσον αφορά τις αποφάσεις που παίρνουμε για να εξαλείψουμε τα, τις στενοπές που υπάρχουν ε, στα κράτη-μέλη θα πρέπει να σκεφτούμε ποια είναι τα μέσα που θα μπορούσαμε να διαθέσουμε στην Ευρώπη για να υπάρχει μια σαφή βάση ιδιών πόρων. Κατά τα άλλα, το θέμα αφορά την παιδεία και την έρευνα και ανάπτυξη, που πολλά μπορούμε να συμβάλλουμε από ευρωπαϊκή πλευρά. Αλλά πάλι το θέμα του οικονομικό είναι αποφασιστικό. έχει το λόγο για 1,5 λεπτό, παρακαλώ. Κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, η πολιτική 2020 στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πάρα πολύ σημαντική για την εξέλιξη της οικονομικής και ε, βιομηχανικής πολιτικής αλλά και της κοινωνικής πολιτικής. Δεν θα πρέπει να ε, προσπαθήσουμε μέσα της πολιτικής αυτής να ε, μειώσουμε όλα τα κοινωνικά δικαιώματα στην Ευρώπη και με σοκάρει το γεγονός ότι η Κομισιόν προ βλέπει μείωση των μισθών και ε, επιδείνωση της κοινωνικής προστασίας. Ορισμένοι συνάδελφοι το ανέφεραν. Οι επιπτώσεις επιτόπου είναι καταστροφικές. Δεν επιτρέπεται οι εργαζόμενοι να είναι εκείνοι που θα πληρώσουν το κόστος της ε, ε, ευρωπαϊκής αυτής παγίωσης. Θα πρέπει να φροντίσουν όλοι να προσαρμοστούν στις εθνικές, στα εθνικά τους δεδομένα για τη νέα πολιτική, γιατί τότε μόνο μπορεί να εξασφαλιστεί η ισορροπία μεταξύ της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης. Τώρα αναφέρονται για τις νέες θέσεις απασχόλησης στα ανοιχτά συμβόλαια. Δεν επιτρέπεται με το να μειώνονται τα δικαιώματα των ε, ε, εργαζομένων να εντάσσονται κατά αυτόν τον τρόπο οι νέοι στην, θέση, στην αγορά απασχόληση, γιατί αυτό οδηγεί μόνο σε επισφαλείς ε, μορφέ εργασία. Οι νέοι είναι εκείνοι που απειλούνται περισσότερο και θα πρέπει να του βοηθήσουμε. Θα πρέπει να μην εργαζόμαστε εκ παραλίλου, αλλά μαζί. Παρακαλώ για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Εγώ αντιλαμβάνομαι το σήμερα και το αύριο ως ότι οι δουλειές θα είναι βιώσιμες ε, μόνο εάν υπάρχει ανταγωνιστική οικονομία και δεν είναι και νομίζω ε, μυστικό για κανέναν ότι υστερούμε στον τομέα αυτό. Για να υπάρχει ανταγωνιστικότητα στην Ευρώπη θα πρέπει να υπάρχει μια θεσμοθετημένη διαδικασία ανταγωνιστικότητας. Θα πρέπει να εντοπίσουμε ποιοι είναι οι παράγοντες της επιτυχίας και να δούμε και πώς θα πρέπει να τους ε, συντεριάξουμε με την κατάσταση. Θεωρώ ότι υπάρχει επαρκής αριθμός ε, μέσων που αφορούν την ανταγωνιστικότητα και ένα επαρκές θεσμικό πλαίσιο το οποίο θα μας επιτρέψει με ελάχιστη πολιτική βούληση να έχουμε μια διαδικασία ανταγωνιστικότητας που θα βασίζεται στο κοινοτικό σύστημα. Εδώ αναφέρομαι στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, ε, την ανάπτυξη που ήδη αναφέρθηκε. Αναφέρομαι και στις ε, διαδικασίες για τις ανισορροπίες, ε, κυρίως για το scoreboard, αυτό το πίνακα αποτελεσμάτων, ο οποίος θα έχει και παράγοντες που σχετίζονται με την ανταγωνιστικότητα. Σχετίζω, αναφέρομαι και στην Ευρώπη του 2020, η οποία θα πρέπει να εφαρμοστεί τώρα και όχι μετά το 2013 και θα πρέπει να υπάρχουν όλες οι πολιτικές ενταγμένες σε αυτήν. Και αναφέρομαι και στην ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής θα πρέπει ε, να ασχοληθούμε όλοι και η αποσύνδεση του πυρήνα τη Ευρώπη από την υπόλοιπη Ευρώπη θα μα οδηγήσει μόνο σε μια διαιρεμένη Ευρώπη. Μπορούμε να έχουμε βιώσιμε θέσει εργασία μόνο αν έχουμε μια ενωμένη Ευρώπη. Μια διαιρεμένη Ευρώπη δεν θα μπορεί να είναι σε καμία περίπτωση ανταγωνιστική Ευρώπη. Για 1,5 λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, σας ευχαριστώ που μου δώσατε το λόγο. Ήμουν η εισηγητής ε, για την έκθεση για τη στρατηγική 2020. Καλωσορίζω την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και συγκεκριμένα του κυρίου Άντρος για το 2011 και τις κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση. Συμφωνούμε και υποστηρίζουμε την πρότασή σας. Προφανέστατα έχουμε τη συνθήκη της Λισαβόνας που σημαίνει ότι ετησίως θα εκπονούμε κατευθυντήριες γραμμές. Εκ του ε, πρέπει να παρακολουθούμε οι αλλαγέ να συνεργαζόμαστε στενά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο και να δούμε αν χρειάζονται κάποιες προσαρμογές. Ως προς τη στρατηγική 2020 ε, θα υπάρξει, θα γίνει αναθεώρηση. Υπάρχει ο θεσμός πλέον του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Οφείλουμε να μεριμνήσουμε ούτως ώστε να ενορθέσει ορθές γραμμέ γραμμές για την απασχόληση, για τα κοινωνικά ζητήματα. Χρειαζόμαστε μύθο τη Αριάδνης για να μπορέσουμε να κάνουμε τις απαιτούμενε προσαρμογές στα αμφιλεγόμενα και προβληματικά ζητήματα, εσχάτως έμαθα ότι τα ε, εθνικά μεταρρυθμιστικά προγράμματα στο παρελθόν έχουν σημειώσει μεγάλες καθυστερήσεις. Ε, δηλαδή, αντί να έχουμε ένα στόχο 100% ε, είχαμε ένα στόχο του 70-72% για την υλοποίηση των κατευθυντήριων γραμμών. Ας προσέξουμε, θυμάστε τις δεσμεύσεις που έχουμε αναλάβει με την στρατηγική της Λισαβόνας, αλλά τελικά δυσκολευτήκαμε πάρα πολύ για την εφαρμογή εφαρμογή ε, Τώρα για του μισθού και τι συντάξει. θα συμφωνήσω μαζί με την Επιτροπή. Ε, έχουμε την αρχή της επικουρικότητας, δεν πρέπει να επεμβαίνουμε υπερβολικά. Εξάλλου έχουμε και εθνικές δεσμεύσεις, τις οποίες πρέπει να τηρήσουμε για τους νέους, για ε, τους ηλικιωμένου, για τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα. Χρειαζόμαστε άλλε ρυθμίσεις.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 30 λεπτά. Ε, αυτό τι είναι. Ευχαριστώ. Ε, δεν νομίζω ότι πρέπει έτσι να ερμηνεύσετε την κατάσταση. Οι συντάξει συνδέονται με την οικονομική υγεία, την ευημερία ενό ε, κράτου. Ε, θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να κατοχυρώσουμε ένα αποτελεσματικότερο σύστημα. Επιθυμούμε ένα ανταγωνιστικό σύστημα, μια ανταγωνιστική και επιτυχημένη Ευρώπη. Αν τα καταφέρουμε, τότε θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε του μη έχοντε σε όσους ε, είναι χαμηλοσυνταξιούχοι, έχουν χαμηλούς μισθούς. Προς το παρόν υπάρχουν σοβαρές διαφορές ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Η κυρία Μόγαν Σαχτιέ για 1,5 λεπτό παρακαλώ. Merci, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Στο πλαίσιο της στρατηγικής 2020, οι κατευθυντήριες αυτές γραμμές της απασχόλησης θα μας βοηθήσουν να αντιμετωπίσουμε τρεις βασικές προκλήσεις. Πρώτον, να εξέλθουμε από την κρίση χάρη στην καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα για να έχουμε μια πραγματική οικονομική ανάπτυξη και έτσι ε, να βοηθήσουμε και την ε, κοινωνία με τα προβλήματά της. Δεύτερον, ε, θα ανανεωθεί μια γενιά ολόκληρη εργαζομένων που συνταξιοδοτούνται τώρα. Τρίτον, θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστική σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία απελευθερώνοντας ε, ε, την οικονομία για τις επιχειρήσεις ε, διότι βαρύνονται από την βαριά φορολογία. Ε, Επίση έχουμε ε, τρει ε, ευάλωτε πληθυσμιακέ ομάδε. Πρώτον, οι νέοι. Πρέπει να αγωνιστούμε γιατί όσοι δεν έχουν δεξιότητες αποκλείονται από την αγορά εργασίας. Να ασχοληθούμε με τους νέου, να διευκολύνουμε την είσοδο τους στην αγορά εργασία, Όχι μόνο με επισφαλείς θέσεις απασχόλησης, όχι μόνο με άσκηση, με στάζ, να καταπολεμήσουμε την ανεργία γιατί είναι χρόνιο πρόβλημα πρόβλημα το οποίο ε, βαρύνει την ε, κοινωνία μας και έχουν ε, πληγεί βαρύτατα από όλους από την κρίση. Δεύτερη ευάλωτη ομάδα, οι γυναίκες επίσης κατέχουν επισφαλίστες απασχόλησης απασχόλησης και χαμηλοαμοιβόμενες. Τρίτον, οι ηλικιωμένοι, οι πιο ηλικιωμένοι πρέπει να διατηρήσουν, διατηρήσουν τη θέση απασχόλησης που έχουν και να χρησιμοποιήσουμε κυρίως το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για να το επιτύχουμε. Ευχαριστώ. Είμαστε στη διαδικασία Catch the έχουν ζητήσει το λόγο πολλοί συνάδελφοι, παραπάνω από είκοσι. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούν να μιλήσουν όλοι. Θα κρατήσουμε την σειρά προτεραιότητα που ζήτησαν το χρόνο και επίσης τους συναδέλφους που ζήτησαν και από την προηγούμενη συζήτηση να παρέχουν και δεν είχαν την ευκαιρία. Λοιπόν, θα δώσω το λόγο πρώτα στον κύριο Σιερ Παρακαλώ. Ένα λεπτό, όχι παραπάνω, κύριε συνάδελφε. Από την παρουσίαση της στρατηγικής Ευρώπης του 2020 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει περάσει περίπου ένα, ένας χρόνος. Δεν ήταν εύκολη η χρονιά αυτή για τα κράτη-μέλη. Τα κράτη-μέλη χρειάστηκαν να καταπολεμήσουν τις συνέπειες της κρίσης. Δράσεις για την εφαρμογή της στρατηγικής ε, ε, έμειναν στο περιθώριο προς το παρόν. Η αύξηση της ε, απασχόλησης, ε, η μείωση των ανθρώπων που ε, βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας και εξελίξεις για την έρευνα και την ανάπτυξη έμειναν όλα αυτά στο περιθώριο και δεν ολοκληρώθηκαν. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν προοπτικές για τη μείωση της ανεργίας που είναι άνω του 10% πανευρωπαϊκά. Αυτό σημαίνει ότι η ανεργία θα είναι υψηλότερη για τα επόμενα χρόνια και επίσης είναι όλο και μεγαλύτερος ο κοινωνικός αποκλεισμός και η ένδυα. Ευχαριστώ. Ένα λεπτό παρακαλώ. Κυρία Πρόεδρε, στον ορίζοντα του 2020, αλλά και πολύ πέρα από αυτή την ημερομηνία, ο συστημικό κίνδυνο που διατρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι να χάσει τη δυνατότητα να είναι ανταγωνιστική ενώπιον των μεγάλων οικονομικών ε, παραγόντων που είναι όλο ένα και πιο εξελιγμένοι τεχνολογικά και όλο ένα και πιο ισχυροί. Η ικανότητα ανταγωνισμού είναι αυτό το οποίο απαιτείται για να αναπτυχθούμε, να αναπτυχθούμε για να δημιουργήσουμε θέσει απασχόληση, να δημιουργήσουμε θέσει απασχόληση και να αναπτυχθούμε για να προστατεύσουμε και να διασφαλίσουμε το κοινωνικό μα μοντέλο. Η μόνη απαραίτητη πρώτη ύλη που διαθέτουμε είναι η γνώση. Και πρέπει να εκμεταλλευτούμε αυτή τη γνώση προκειμένου να καινοτομήσουμε, να προσαρμοστούμε στι αλλαγέ, αλλά και να είμαστε επικεφαλεί αυτών των αλλαγών. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να επενδύσουμε ακόμα περισσότερο σε πανεπιστήμια, στο εκπαιδευτικό μας σύστημα, στην έρευνα και στην ανάπτυξη, προκειμένου να γίνουμε μία δύναμη σε αυτό το οποίο μπορούμε να είμαστε δύναμη, στη γνώση. θα πάρει το λόγο. Ένα λεπτό παρακαλώ. Arvoisa puheenjohtaja, arvoisa komission jäsen, nämä tavoitteet Eurooppa 2020 Κύριε Επίτροπε, κύριε Πρόεδρε, οι στόχοι της Ευρώπης 2020 είναι πολύ φιλόδοξη και θα ήθελα να εκμεταλλευτώ αυτό το χρόνο αγόρευσης που έχω για να δούμε τι πρέπει να κάνουμε στην πράξη προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί και να μην αποτύχει η στρατηγική μας. Παραδείγματος χάρη, θα πρέπει σε όλη την Ευρώπη να εξετάσουμε τις περιφέρειες. Δεν μπορούμε να έχουμε μια προσέγγιση για όλους. Ε, το συζητήσαμε αυτό και χθε και θα πρέπει να σκεφτούμε την πολιτική συνοχή και να την εκμεταλλευτούμε ώστε να υπάρχουν περισσότερε θέσει απασχόληση, περισσότερη καινοτομία και για να γίνει αυτό χρειαζόμαστε μια πολιτική που θα καλύπτει όλη την Ευρώπη ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί αναπεριοχή. Θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να έχουμε χρήματα για τους τομείς αυτούς, αλλά καταρχάς χρειαζόμαστε μια πολιτική που να είναι αποτελεσματική. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Υπάρχουν ε, αυτά τα προβλήματα εδώ και πολύ καιρό και δεν λαμβάνονται υπόψη στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, μεταξύ αυτών είναι όλες οι, υπάρχουν όλες οι κοινωνικές επιπτώσεις τόσο αρνητικές για τους πολίτες. Εάν το δούμε εν των 25 εκατομμυρίων ε, ανέργων, των εκατομμυρίων εργαζομένων που πληρώνονται άσχημα 85 εκατομμύρια που ζουν σε συνθήκες φτώχειας. Ε, ε, βλέπουμε ότι αυξάνονται συνεχώς, οξύνονται τα προβλήματα. Μα είμαστε απειβδισμένοι. με τις κοινωνικές ρυθμίσεις δεν φροντίζουμε τους πολίτες και βλέπουμε ότι εκατομμύρια ανέργων ε, γυναίκες, ε, νέοι θέλουν ε, να καταπολεμήσουν τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εμείς μιλάμε για το σύμφωνο της ανταγωνιστικότητας και άλλα τέτοια παρεμφερή. Πρέπει να σεβόμαστε τους ανθρώπους, να σεβόμαστε τους μισθωτούς. Εγώ τώρα θα πάρει ένα λεπτό παρακαλώ. Κύριος Ρώση. Αξιότιμοι συνάδελφοι, συμφωνώ ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να έχει χρόνο στη διάθεσή του ώστε να προτείνει τις καλύτερες πολιτικές για την απασχόληση για το 2020. Επειδή βιώνουμε αυτή την κρίση που βιώνουμε στην Ευρώπη, δεν μπορούμε να παραμελήσουμε και τις ανάγκες των πολιτών είναι απαραίτητο να προβλέψουμε βοήθεια στις οικογένειες, τους νέους που ψάχνουν μια θέση εργασίας και όλοι, ε, όλους όσους βρίσκονται άνεργοι μετά από μια μακρά ε, επαγγελματική σταδιοδρομία. Θα πρέπει να διασφαλίσουμε λοιπόν πρώτα την εργασία για τους πολίτες μας και μετά για τους υπολείπους. Θα πρέπει να υπάρχει συντονισμός μεταξύ των ε, γραφείων εξέβρεσης εργασίας στην Ευρώπη ώστε να μπορέσουν να γνωρίζουν όλοι στην Ευρώπη ποιες είναι οι θέσεις εργασίας που είναι διαθέσιμες. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει υπάρχει προστασία στα σύνορα για να υπάρχει ανεξέλεγκτη εισβολή από τις χιλιάδες μετανάστες που λόγω της κατάστασης του Μαγκρέμπ θα εισβάλλουν στις, ε, στα εδάφη μας. Μόνο οι ελεγχόμενες ε, θέσεις εργασίας για τους πολίτες μας ε, θα αποτρέψουν την εισβολή πολιτών από τρίτες χώρες και δεν θα έχουμε ανάπτυξη και κοινωνική ανάπτυξη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όσον αφορά την στρατηγική, οι προσδοκίε είναι διαφορετικέ. Οι μεν περιμένουν ότι εδώ δεν κάνουμε τίποτα και ότι η στρατηγική αυτή δεν αξίζει το χαρτί πάνω στο οποίο έχει τυπωθεί. Απ' την άλλη μεριά βλέπουμε πραγματικέ προκλήσεις που να έρχονται να τι αντιμετωπίσουμε. Το αποτέλεσμα είναι ότι βλέπουμε εδώ μεταξύ άλλων και dumping μισθολογικό. Η στρατηγική θα πρέπει να είναι ε, ότι θα πρέπει το 40% λέμε μιας γενιάς να έχουν δίπλωμα πανεπιστημίου. Προς τι? Προς τι? Βλέπετε τι γίνεται στην Ιταλία όπου υπάρχουν εκατομμύρια αποφύτων πανεπιστημίων που δεν έχουν τις κατάλληλες θέσεις εργασίας. Νομίζω ότι αυτό που χρειαζόμαστε είναι καλύτερη κατάρτιση επαγγελματική, ναι, αλλά δεν θα το πετύχουμε αυτό εάν το 20% του πληθυσμού έχει ένα δίπλωμα από το Πανεπιστήμιο. Αυτό δεν είναι σωστή άγουσα. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ράγχελ το λόγο θα πάρει τώρα. <coughs> Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να καταγραφεί ότι είναι θεμελιώδες ε, και το τονίζω στην εποχή αυτής της οικονομικής κρίσης ναι, να επενδύσουμε στην οικονομική ανάπτυξη και στις αναπτυξιακές στρατηγικές. Χρειαζόμαστε επίσης μια ε, κρατεά πολιτική απασχόλησης. Εάν έχουμε μια σωστή τέτοια πολιτική θα λύσουμε το οικονομικό πρόβλημα αλλά και το κοινωνικό. Θα ήθελα λοιπόν να περάσω ένα μήνυμα για να ληφθεί υπόψη στη στρατηγική 2020 για ένα κομμάτι του πληθυσμού, για τους νέους ή έχουν Μεγάλη βαρύτητα. Το ίδιο και οι ηλικιωμένοι. Πάνω από τα 50 χρόνια προσεγγίζουν την συνταξιοδότησή τους και πρέπει να τους φροντίσουμε. Αν θέλουμε να βελτιωθεί η κατάσταση πρέπει να καταπολεμήσουμε τις επισφαλείς θέσεις απασχόλησης για τους άνω των 50 ετών. Σίλα, θα πάρει το λόγο τώρα. Ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε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 θεωρώ ότι για την απασχόληση θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε τα μοντέλα απασχόλησης που έχουμε στη διάθεσή μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να στηρίξουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και να αποτιμήσουμε το δυναμικό τους για να δημιουργήσουμε νέες θέσει απασχόλησης μεταξύ των στόχων μας, των αναπτυξιακών μας στόχων. Ε, ε, είναι και η καταπολέμηση της φτώχεια ε, και θα πρέπει να αποδίδουμε ιδιαίτερη βαρύτητα όλα τα σκέλη τη στρατηγική ε, για να έχουμε μια οικονομική ανεξαρτησία στρατηγική 2020 ε, οφείλει να είναι υποφελής για όλους τους πολίτες. Ε, για να γίνει αυτό όλοι θα πρέπει να υπομιστούν τις δικές τους ευθύνες, δηλαδή σε τοπικό, σε περιφερειακό, σε εθνικό επίπεδο. Ευχαριστώ. Έχει το λόγο παρακαλώ. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Οι κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση θα πρέπει να θεωρούνται βασικό εργαλείο για την ε, διαχείριση της μακροπρόθεσμης ανάπτυξης και αυτό ε, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Οι κατευθυντήριες γραμμές είναι το μέσο μέσω των οποίων τα κράτη-μέλη θα μπορέσουν να έχουν εθνικές μεταρρυθμίσεις. Και η επιτυχία της στρατηγικής ε, για την Ευρώπη 2020 συνδέεται άρρηκτα με αυτό τα προγράμματα μεταρρύθμισης θα πρέπει να εφαρμοστούν μέχρι τον Απρίλιο. Αναφέρομαι επίση και στην Επιτροπή των Περιφερειών και θα ήθελα να επισημάνω πόσο σημαντικό είναι να συμμετέχουν και οι περιφέρειε σε αυτό το έργο. Το να γίνουν αλλαγέ αυτή τη στιγμή θα μπορούσε να αποσταθεροποιήσει τη διαδικασία. Παρακαλώ λοιπόν σημειώστε ότι χρειαζόμαστε μια οριζόντια προσέγγιση για την εφαρμογή τη στρατηγική τη Ευρώπη 2020. Επαναλαμβάνω λοιπόν για άλλη μια φορά πόσο σημαντική είναι η πολιτική συνοχή για την Ευρώπη του 2020. Ďakujem pekne pani predsednička, pán komisár. Štyri usmernenia Rady pre politiky... Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Τέσσερις κατευθυντήρες γραμμές θα πρέπει να διέπουν την εργασία μας και το έτος 2011. Δεν θα πρέπει να τις παραβλέψουμε. σύμφωνα με την αρχή της ε, ζήτησης και της προσφοράς πρέπει να κινηθούμε. Αυτό ε, λειτουργεί πολύ καλά. Η αύξηση της, ε, των ικανοτήτων εργασίας των γυναικών είναι πάρα πολύ σημαντική. Θα πρέπει τα κράτη-μέλη να αναγνωρίσουν από την άλλη μεριά την εργασία των μητέρων και τη συμβολή που προσφέρουν στο ΑΕΠ. Το κράτος θα έπρεπε να συγκεντρώσει την προσοχή του στην, ε, στην καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, γιατί είναι πολύ δύσκολο να βρει από αυτή την ε, παγίδα. Κυρία Μπέρες, Έχετε το λόγο, εσύ, κυρία Σίγητρια. Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ τον Επίτροπο μπορείτε να πείτε στον πρόεδρο Μπαρόζο ότι πολύ θα θέλαμε να είχε έρθει να συμμετάσχει σε αυτή τη συζήτηση. Είναι η πρώτη που γίνεται για τις ε, ε, προκλήσεις σχετικά με την ετήσια εξέταση των καθηγητριών γραμμών απασχόλησης, δηλαδή τον ακρογωνιαίο λίθο ε, του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου το, που, είναι, που του είναι τόσο προσφυλές. Επίσης, υπό αυτές τις προϋποθέσεις δεν θα είμαστε εύκολοι στη συνεργασία μας να το ξέρετε το οικονομικό οικονομικό πακέτο συνεπάγεται ότι, μάλλον για να εγκριθεί, συνεπάγεται ότι θα ε, αποδώσει μεγαλύτερη βαρύτητα σε αυτά που λέμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πιστεύει ότι πρέπει να εφαρμοστεί ολόκληρη η συνθήκη τη Λισαβόνα και συγκεκριμένα το άρθρο 9 που προβλέπει ότι το τα κοινωνικά ζητήματα είναι οριζόντια ζητήματα. Δεν θέλουμε να μείνει κενό γράμμα αυτό το άρθρο. Ε, επιμένουμε, διεκδικούμε την πλήρη εφαρμογή τη συνθήκη. Ε, σχετικά με την ελάχιστη αναθεώρηση της συνθήκης, ε, κοιτάξτε, πρέπει να εκμεταλλευτούμε πριν να αναθεωρήσουμε όλο το δυναμικό της υφιστάμενης συνθήκης και συγκεκριμένα το άρθρο 9 για τα κοινωνικά ζητήματα. Ε, να σα πω τι μου έκανε εντύπωση στη σημερινή μα συζήτηση. Έχουμε ορισμένε φορέ την εντύπωση ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρά την κρίση συνεχίζει να ε, ε στοχάζεται επί τη βάση των παλαιών συνταγών, των παλαιών λύσεων. Για την αγορά εργασίας όμως, ε, ε, όταν μιλάμε για τη μεταρρύθμιση της αγοράς εργασίας, ε, όλοι μιλάνε για την ευελιξία, όχι για την ευελιξία ασφάλεια, για την ευελιξία. Αλλά την προηγούμενη δεκαετία, πριν εκδηλωθεί μάλλον η κρίση, επικρατούσε η ιδέα ότι αρκεί η ανάπτυξη για να έχουμε θέσει απασχόλησης. Μα δεν επαρκεί αυτό. Ποιο είναι το πραγματικό διακύβημα, η πραγματική πρόκληση, η απασχόληση. Και για μας και για τις χώρες που περιβάλλουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βλέποντας όμως τη συζήτηση που γίνεται για την ανταγωνιστικότητα, διαπιστώνω ότι δεν ε, γυρνάμε την πλάτη ουσιαστικά στην προτεραιότητα της απασχόλησης και ανησυχώ. Τώρα το λόγο θα πάρει ο Επίτροπος ο κύριος Σάντορ, εξ ονόματος Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχετε το λόγο κύριε Επίτροπε. Thank you much. Uh, ε, ευχαριστώ Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτές. Ε, με εμπνέει η σημερινή συζήτηση, ε, τροφοδοτεί τον προβληματισμό μας. Ε, ήγηραν οι συνάδελφοι πολύτιμα σχόλια, εύστοχες παρατηρήσεις για την ετήσια έκθεση, για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και γενικότερα για τη στρατηγική 2020. Το σημαντικό είναι να έχουμε μια σαφή εικόνα και για την οικονομική κατάσταση και τα στοιχεία που έχουμε στα διάθεσή μας. Η αλήθεια, αν και δεν μας βολεύει είναι ότι ε, ε, ανακάμπτει οικονομικά η Ευρώπη. Ήδη από πέρσι είχαμε ε, ανάπτυξη, όχι σε όλα τα κράτη-μέλη. Ε, και το δεύτερο που δεν βολεύει κάποιους είναι ότι ε, ε, υπάρχει μεγά, υπάρχουν μεγάλες διαφορές ανάμεσα στα κράτη-μέλη και είναι αδύναμη αυτή η οικονομική ανάκαμψη. Οπότε πρέπει να προσαρμόσουμε ανάλογα τις πολιτικές μας, να διατηρήσουμε αυτή τη δυναμική της ε, οικονομικής ανάκαμψης ε, ε, και να διορθώσουμε αυτές τις ανισότητες στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πλην όμως δεν είναι αυτό εφικτό εάν δεν διορθώσουμε τις αδυναμίες που κατέστησαν σαφείς με την κρίση και να βελτιώσουμε την, το μοντέλο οικονομικής διακυβέρνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εδώ αρχίζει να περιπλέκεται η υπόθεση διότι ε, αληθεύει ότι δεν αναγνωρίζουν όλοι αμέσως ε, όλες οι προτεραιότητες. Ε, για μας η προτεραιότητα είναι η ανάπτυξη και όλες οι υπόλοιπες πολιτικές σε αυτό το στάδιο εξυπηρετούν αυτόν τον στόχο πρέπει να τονώσουμε την ανάπτυξη, να γίνει ισχυρότερη, κρατεότερη ανάπτυξη και για να γίνει αυτό χρειαζόμαστε ένα αυξημένο επίπεδο χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και εξυγίανσης των δημοσιοοικονομικών. Είναι αναπεόφευκτο για τα επόμενα χρόνια. Δηλαδή, δημοσιονομικός, η η δημοσιονομική εξυγίανση θα συνεχίσει να μας απασχολεί τα επόμενα χρόνια και έτσι ε, θα είναι συνεκτική η πολιτική μας σχετικά με την ε, κυκλική παρέμβαση που χρησιμοποίησαν ε, τα κράτη-μέλη για να το αντιμετωπίσουν την ύφεση τα τελευταία χρόνια. Δημοσιονομική εξυγίανση λοιπόν, η οποία όμως δεν θα πλήξει την ζήτηση, ε, δεν θα πλήξει την οικονομία. Ε, μια ευφυή εξυγίανση χρειαζόμαστε που θα ε, διατηρήσει την ακαιρεότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας εν γέννη. Πρέπει να μάθουμε αυτό το μάθημα, χρειάζεται σταθεροποίηση, θα μπορούσα βέβαια να χρησιμοποιήσω και άλλη φρασιολογία, αλλά ε, δεν θα το κάνω. Ε, πρέπει να σταθεροποιήσουμε το ευρώ, την νομισματική ένωση. Ε, και για να γίνει αυτό θα πρέπει να τονίσουμε το οικονομικό σκέλος αυτής της ένωσης, το συντονισμό δηλαδή των οικονομικών πολιτικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα ήθελα να θέσω ένα ρητορικό ερώτημα η ενίσχυση του οικονομικού σκέλους ε, της διακυβέρνησης μπορεί να επιτύχει εάν δεν ε, συνεργαστούμε περισσότερο σχετικά με την ε, μισθοδοσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί το λέω αυτό. Στην αιτήσια δημοσκόπηση, ε, μάλλον έρευνα για την οικονομία, δεν ετονίζεται ίσως επαρκώς, ε, μας είπατε, η σημασία του κοινωνικού διαλόγου. Μα το αντίθετο, στις χώρες όπου υπάρχει ε, μακρά παράδοση κοινωνικού διαλόγου, βλέπουμε ότι διέρχονται από την κρίση με λιγότερες απώλειες ως προς τους ανθρώπινους πόρους. Έχει παραμείνει σε χαμηλότερα επίπεδα η ανεργία σε αυτά τα κράτη-μέλη και γι' αυτό προτείνουμε την ενίσχυση του κοινωνικού διαλόγου σε κράτη που υπέφεραν περισσότερα από την κρίση γιατί ε, έδωσαν ε, μια λιγότερο ευέλικτη αν θέλετε απάντηση ε, στην κρίση όπως η Ολλανδία, η Αυστρία και η Γερμανία. Ε, να αυξήσουμε λοιπόν, ε, να αναβαθμίσουμε το κοινωνικό διάλογο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, το διάλογο δηλαδή που κάνουμε με τους ε, κοινωνικούς εταίρους. Το Μάρτιο έχουμε ε, διοργανώσει ήδη το φόρουμ με τους ε, κοινωνικούς εταίρους για να ενισχύσουμε αυτόν τον διάλογο. απορρίπτω κατηγορηματικά την ιδέα ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεχίζει να μην συνέβαινε τίποτα. Όχι. το πέρσι, από πέρσι έχουμε δρομολογήσει διάφορες ε, ε, ποιοτικές ε, πρωτοβουλίες. Ενίσχυση του χρηματοπιστωτικού κανονισμού. Μην υποτιμούμε την εργασία του Επιτροπού Μπαρνιέ. Για τη στρατηγική 2020 παρουσιάσαμε μια νέα βιομηχανική πολιτική σε ευρωπαϊκό επίπεδο που δίνει ιδιαίτερη σημασία στην ανταγωνιστικότητα και στην βιωσιμότητα των θέσεων απασχόλησης στην Ένωση. Επίσης, ε, ρηξικέλευθες προσεγγίσεις μας βοηθούν να τονώσουμε τις επενδύσεις και να βρούμε και την χρηματοδότηση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται για να, ε, διαρκώς για να εκπονεί καινοτόμα χρηματοδοτικά μέσα ε, ένα θα αφιερωθεί στην ε, ε, αναβάθμιση των ενεργειακών δικτύων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι απαραίτητο αυτό για να αναπτυχθεί η ενεργειακή αγορά. Χρειαζόμαστε λοιπόν την απαιτούμενη υποδομή. Είναι κέρια σημασία. Επίσης, το μέσο της μικροχρηματοδότησης ε, να ευχαριστήσω το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την συγκατάθεσή τους πέρσι ε, και στην ε, Ολλανδία ξεκίνησε ε, να λειτουργεί το μέσο μικροχρηματοδότησης ε, και έπονται και άλλα έτσι ε, κάποιοι άνεργοι θα μπορέσουν να δραστηριοποιηθούν και πάλι στην αγορά εργασίας μπορούν να γίνουν επιχειρηματίες ή κάποιοι που ήδη εργάζονται ναι, μπορεί να θέλουν να ανακυκλωθούν ή μπορεί να θέλουν να αλλάξουν κατεύθυνση μετά τα 50 τους, μετά τα 60 τους, γιατί όχι συζητούμε τι ε, στρατηγικέ ε, απασχόλησει. Την περασμένη εβδομάδα στο Συμβούλιο ΕΠΣΚΟ στο Κούντελη, στην Ουγγαρία συζητήσαμε ε, το πώ θα μπορούσαμε ναι, να δημιουργήσουμε και άλλε θέσει απασχόλησης και κυρίως πώ να βοηθήσουμε τι πληθυσμιακέ ομάδε που είναι και στη δυσαιρέστερη θέση. Δυστυχώ του νέου ενώ σε κάποια κράτη-μέλη είναι τραγική η κατάσταση και τονίζω ότι υπάρχουν σοβαρέ διαφορέ ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Σε κάποια ε, η ανεργία ευτυχώ είναι σε σχετικά χαμηλά επίπεδα, αλλά ο μέσο όρο Ευρωπαϊκή Ένωση είναι υψηλό ε, Σε βαλτικέ ε, Ισπανία, παραδείγματος χάρη, είναι καταστροφική η στην ισπανια παραδειγματο ειναι καταστροφικη η κατασταση και έχουμε προειδοποιήσει της κυβερνήσεις αλλά χρειάζεται ένα περίπλοκο μείγμα πολιτικών για να το αντιμετωπίσουμε για την παιδεία, για την απασχόληση, άλλου είδους μέτρα για να διορθώσουμε την κατάσταση. Αλλά δεν είναι μόνο αυτή η προβληματική ομάδα. Έχουμε ε, άλλες ε, δύο γυναίκες εκεί ηλικιωμένοι και γι' αυτό ε, ξεκινήσαμε και το Ευρωπαϊκό Έτος ε, για τους ηλικιωμένους σχετικά με τις ερωτήσεις σας τώρα για τις κατευθυντήριες γραμμές απασχόλησης πιστεύω ότι όλοι συνεχίζουμε να εστιάζουμε σε αυτές για να γίνει πιο ουσιαστικό το περιεχόμενό του. Ε, στο άρθρο 148 τη συνθήκη προβλέπεται σαφή ρόλο για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, και θα ε, επαναληφθούν οι κατευθυντήριε γραμμέ απασχόληση, θα επαναβεβαιωθούν. Τι σημαίνει αυτό. Θέλουμε να συνεχίσουμε και το 2014 να είναι σταθερέ και να μην υπερσκελίζονται από την ετήσια έρευνα. Να, Δηλαδή οι κατευθυντηρίες ε, γραμμές είναι πιο μακροπρόθεσμες, ε, η αιτήσια έρευνα είναι αιτήσια. Ε, αληθεύει επίσης ε, ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνεται αυτή η ετήσια έρευνα και αποδίδει μια σημασία στη στρατηγική 2020 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, θα εμπλακεί με διάφορους τρόπους ε, στις εργασίες και τις συζητήσει. Ε, θα αναφερθώ στο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, στις σχετικές διαπραγματεύσεις, το προϋπολογισμό προφανώς που θα απηχεί τις προτεραιότητες της στρατηγικής 2020 και προφανώς θα ενημερώνεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την εκπόνηση των εθνικών μεταρρυθμιστικών προγραμμάτων καθώς και των συστάσεων κάθε, προς κάθε μεμονωμένο κράτος μέλος σαφές ε, ότι εξ αρχής υπάρχει ανησυχία για το μέλλον της στρατηγικής 2020. Ένα φάσμα στοιχιώνει την ε, στρατηγική του 2020. Ποιο είναι αυτό η στρατηγική της Λισαβόνας. Ε. Εδώ στο Κοινοβούλιο επανειλημμένα έχουμε συζητήσει μαζί γιατί πιστεύουμε ότι θα έχει περισσότερη επιτυχία, μεγαλύτερη επιτυχία μάλλον η στρατηγική 2020 γιατί έχει πιο συγκεκριμένους στόχους σε σχέση με τη στρατηγική της Λισαβόνας. Νομίζω ότι μόνο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να εξασφαλίσει ότι θα υπάρξει κάποια συνοχή ανάμεσα στις διάφορες ε, πρωτοβουλίες. Ε, ε, θα ε, έχουμε διάφορα στοιχεία όπως η ενιαία αγορά, η πολιτική συνοχή, η πολιτική απασχόληση, η διαθροτική πολιτική, όλα αυτά συναποτελούν ε, την γενικότερη οικονομική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η βαρύτητα θα πρέπει να αποδώσουμε σε όλα αυτά τα επιμέρους στοιχεία και προφανώς εμείς δεν θέλουμε να οικοδομήσουμε μια Ευρώπη δύο ταχυτήτων ε, και πρέπει να ε, προσέξουμε ούτω ώστε να μην υπάρξει πολιτικό διχασμός λόγω των ανισοτήτων προ την οικονομική ανάπτυξη. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους εσάς που συμβάλλατε πολύ υποκοδημητικά σε αυτή τη τόσο χρήσιμη συζήτηση. Θα ήθελα επίση να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την κυρία Μπερές για τη θαυμάσια έκθεσή τη. και τις πολύ σημαντικές παρατηρήσεις και κριτικές που εκφράζει. Ίσως ε, διαφορετικά εκτιμούμε την πραγματικότητα, όπως είπατε και όπως είπε και η κυρία Βούγνα, και όσον αφορά την κρίση και όσον αφορά την ανάκαμψη. Αλλά πιστεύω ότι συμφωνούμε όλοι πάνω σε ένα σημείο ότι κανένας δεν θέλει να υπάρχει ανάκαμψη χωρίς απασχόληση και όλοι προσπαθούμε να επιτευχθεί η ισορροπία μεταξύ της φορολογικής παγίωσης και της ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης. Η δημοσιονομική πειθαρχία και η ανάπτυξη της απασχόλησης θα πρέπει να προχωρούν από κοινού. Ε, Έχω κάτι πιο γενικό να πω όσον αφορά τα οικονομικά θέματα. Ξέρουμε ότι έχουμε τώρα μία ε, πλήρη δέσμη, πλήρη προσέγγιση μια συνολική δέσμη θα μπορούσαμε να πούμε, εκ των οποίων τα περισσότερα στοιχεία αναφέρθηκαν από τον Επίτροπο Και θα ήθελα να τονίσω ότι θα πρέπει να συγκεντρώσουμε την προσοχή μας σε δύο από τα στοιχεία αυτά τις δέσμες. Το ένα, η εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Πρώτη φορά γίνεται κάτι τέτοιο. Θα έχει σημαντική επίπτωση στις μελλοντικές εξελίξεις της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Δύο θα ήθελα να φέρω εδώ. Καταρχήν, το χρονοδιάγραμμα είναι πολύ στενό, θα πρέπει να σεβαστούμε λοιπόν όλοι τις προθεσμίες. Και δεύτερον, υπάρχουν στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν και θα πρέπει να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια ούτω ώστε το, συνολικό, το σύνολο συγγνώμη, των προθεσμιών να τηρούνται από κάθε ένα κράτος μέλος. Όσον αφορά την απασχόληση και την καινοτομία και για την ενέργεια βέβαια, θα ήθελα να πω για την ενέργεια, ότι η Λαβέ χώρα μια πολύ σημαντική συνάντηση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 4 Φεβρουαρίου, που για πολλούς ε, αποτελούσε ένα ορόσημο και για την δημιουργία της ολοκληρωμένης αγοράς ενέργειας και για την αποτελεσματική χρήση ενέργειας και όσον αφορά τις εξωτερικές πτυχές της κοινή ενεργειακής πολιτικής. Ε, για όλα αυτά τα σημεία λήφθησαν πολύ σημαντικές αποφάσεις. Και, τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό, θα ήθελα να αναφερθώ στην καταπολέμηση της ένδυας, στην καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και εδώ θα ήθελα να αναφερθώ στο ψήφισμα το οποίο μόλις ε, υιοθετήσατε όσον αφορά την ενσωμάτωση των Ρωμά. Θα ήθελα να σας χαρώ και να ευχαριστήσω τον Ιαροκορίδιο που έπαιξε αποφασιστικό ρόλο στην προετοιμασία της έκθεσης αυτής και στην υιοθέτηση αυτού του τόσο σημαντικού ψηφίσματος. Θα ήταν πολύ χρήσιμο για μας. Θα είναι το έγγραφο αυτό πολύ χρήσιμο για μας όταν εργαστούμε και προετοιμάσουμε το πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την ένταξη των Ρωμά. Το άλλο θέμα που θα ήθελα να σας μιλήσω τώρα είναι τα έξι νομοθετικά κείμενα που υπάρχουν εδώ και θέλω να διαβεβαιώσω την κυρία Σλεπικουράν ότι δεν θέλουμε μόνο να ακούσουμε το Κοινοβούλιο αλλά θέλουμε και πρέπει να συμφωνήσουμε μαζί του υπό τους όρους της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας. Θα πρέπει να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια ώστε αυτή η διαδικασία να επιταχυνθεί και να ολοκληρωθεί επιτυχώς μέχρι τα τέλη της Ουγγρικής Προεδρίας. Δεν θέλω να επισέλθω σε όλα τα άλλα στοιχεία τη δέσμη αυτή, αλλά ένα πράγμα θα ήθελα να τονίσω. Το Συμβούλιο θέλει να σεβαστεί πλήρω την κοινοτική μέθοδο. Δεν έχουμε καμία επιφύλαξη πάνω σε αυτό το θέμα. Όπως είπαμε και στο παρελθόν, η συνθήκη τη Λισαβόνα πολλά άλλαξε. Υπάρχουν σημαντικέ αλλαγές, των οποίων τι επιπτώσει γνωρίζουμε όλοι, αλλά η συνθήκη της Αβώνας δεν άλλαξε την καρδιά της ευρωπαϊκής δομής και αυτό είναι η, κοινωνική, η κοινωτική μέθοδος. Βέβαια, πάντα πρέπει να ευθυγραμμιστούμε με τη συνθήκη, οτιδήποτε και αν κάνουμε. Και θα ήθελα να σα τονίσω ότι αν διαβάσει κανένα προσεκτικά τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τη 4 η Φεβρουαρίου θα δείτε ότι οτιδήποτε, οτιδήποτε λέγεται εκεί πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένο με τη συνθήκη. Το τελευταίο μου σχόλιο θα είναι πολύ σύντομο. Για τα χρήματα. Όπως είπε η κυρία Λένα Εκ, όλες αυτές οι πολιτικές χρειάζονται χρήματα, χρειάζονται χρηματοδότηση. Οπωσδήποτε συμφωνώ μαζί σας. Αλλά υπάρχουν διαφορές. Υπάρχουν διαφορές λέγω την προσέγγιση των κρατών μελών. Αυτή τη στιγμή θα ήθελα να τονίσω ένα πράγμα από σκοπιάς προεδρίας. Συστήνουμε πρώτα να συζητήσουμε την ουσία και μετά να συζητήσουμε χρήματα, αριθμούς και πόρους. Θα είναι μακρά η συζήτηση, έχουμε χρήσιμες συζητήσεις προσανατολισμού για την πολιτική συνοχής, ε, ενέργειας, γεωργίας και ούτω καθεξής. αλλά δεν επιτρέπεται όπως λένε να ξεκινήσουμε από το τέλος σε γενικές γραμμές λοιπόν θα θέλαμε να βοηθήσουμε σε όλες αυτές τις συζητήσεις και να καταλήγουμε στην πραγματική, στην τελική συζήτηση για τους πόρους. Για άλλη μια φορά θα ήθελα να συγχαρώ όλους εσάς και να σας ευχαριστώ για τη συζήτηση. Κυρίες Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η κοινή συζήτηση έληξε. Έχω λάβει έξι προτάσεις ψηφίσματος για το θέμα της συζήτησης σχετικά με την Ευρώπη 2020 και μία πρόταση ψηφίσματος για το θέμα της συζήτησης σχετικά με την πολιτική των κρατών μελών στον τομέα της απασχόλησης. Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί αύριο στις 12 το μεσημέρι για τα θέματα αυτά που μόλις συζητήσαμε. Έχει διαδικαστικό ο κύριο Οντί. Παρακαλώ, Monsieur Οντί, vous avez, vous avez ε, ε, question de motion d'ordre. Madame Πρόεδρε, δικαίω ο κύριος Υπουργό αναφέρθηκε στο σεβασμό της συνθήκης, Αλλά τόνισε ότι υπήρξε ένα Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 4 Φεβρουαρίου. Θα ήθελα, εφαρμόζοντας το άρθρο 15 της συνθήκη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πότε ο πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα έρθει να μας παρουσιάσει τα αποτελέσματα του Ευρωπαϊκού αυτού Συμβουλίου ενώπιν του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Γιατί δεν θα έρθει νομίζω αυτή η σύνοδο. Το σημειώνουμε. Ευχαριστούμε. Και